Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Καλημέρα σε όλους. Θα ξεκινήσουμε με το σημείο 20. Ε, η ενδιάμεση συμφωνία για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027. Έχουμε προετοιμάσει ε, ε, στη ε, γνωμοδότηση συγγνώμη, για την αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή που είναι η Επιτροπή Προϋπολογισμού θα δώσω το λόγο στον συνάδελφο για πέντε λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, ε, η γνωμοδότηση αυτή μας δίνει την ε, δυνατότητα να δώσουμε τη δική μας άποψη στην Επιτροπή Προϋπολογισμών αλλά και στην, Επιτροπή, ε, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την άποψή μας για το πολιετές δημοσιονομικό πρόσιο. Θα ήθελα να σας πω ότι το, αυτό το πει πρέπει να αποτελέσει το πολιετές, πολιετές πρόγραμμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση όπου θα αναφέρονται όλες οι προτεραιότητα στο έγγραφο είναι, ε, είναι ε, σύντομο γιατί ξέρετε ότι υπάρχουν ε, κάποιοι περιορισμοί όσον αφορά το μέγεθος μιας γνωμοδότησης. Και γι' αυτό κάναμε μια προσπάθεια να περιλάβουμε εδώ όλα τα στοιχεία τα οποία θα έπρεπε οπωσδήποτε να αναφερθούν ως ορόσημα θα ήθελα να προτείνω αυτή τη φορά ε, να ενδιαφερθούμε για θέματα, ε, σε θέματα εμπορικής ε, πολιτικής καθώς επίσης σε συμφωνίες σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο. Οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών θα πρέπει να αποτελέσουν πλέον το ορόσημο όσον αφορά και τα προτιμησιακά καθεστώτα και την εμπορική ε, πολιτική. Η περίοδος 21-27 θα είναι αποφασιστική σημασία έτσι ώστε ο πλανήτης να μπορέσει να επιτύχει ε, τους ε, στόχους αυτούς. Βεβαίως πολλές αλλαγές θα προκύψουν και πρέπει να σας πω ότι ε, δεν ξέρω εάν είναι σωστό να δημιουργήσουμε αυτό το τεράστιο ε, εργαλείο το οποίο ίσως θα έχει σαν αποτέλεσμα ε, την μείωση της εστίασης που είναι τόσο σημαντική για την χρηματοδότηση της ανάπτυξης. οπωσδήποτε πάντως ε, θα γίνει και μία ε, έκθεση η οποία θα είναι αφιερωμένη ακριβώς σε αυτό το θέμα. Σίγουρα όμως θα πρέπει να υπάρξει η απαραίτητη ευελιξία έτσι ώστε ε, να χρηματοδοτηθούν όλες και θα πρέπει οπωσδήποτε αυτό να συνεχιστεί και στο μέλλον έτσι ώστε να μπορέσουν να χρηματοδοτηθούν όλες οι εταιρικέ σχέσεις και όλες οι σχέσεις μας με τις χώρες εταίρους γιατί οι χώρες αυτές χρειάζονται και τη βοήθειά αλλά είναι και σημαντικές ε, και για μας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να προωθήσουμε σωστά τις εμπορικές μας συμφωνίες βάσει των νέων, ε, της νέας πραγματικότητας. Ε, επίσης θα πρέπει να δούμε ε, ποια είναι η ε, επίπτωση στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων, στην οικονομική, την κοινωνική ζωή των ανθρώπων, ποια είναι η επίπτωση, λέω, των εμπορικών μας συμφωνιών, εάν είναι δυνατόν να αναπτυχθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εδώ συμπαραλαμβάνονται και, κάποιες, και κάποια πολύ περίπλοκα στοιχεία παραλλήλων, σωρευτικά, παραλλήλων συμφωνιών ή ε, πρωτοκόλων ε, έτσι ώστε ε, να ε, ε, δούμε στοιχεία τα οποία μπορούν να βελτιώσουν την ε, αποδοτικότητα. Έχουμε την δυνατότητα να βελτιώσουμε τις συμφωνίες μας έτσι, και, έτσι ώστε να βελτιώσουμε γενικότερα την κατάσταση όσον αφορά τώρα την απώλεια εισοδημάτων λόγω δασμολογικών φραγμών. Θα πρέπει η Κομισιόν να δώσει τα ακριβή ποσά και οπωσδήποτε να επιτηρεί το, το σύστημα των δασμών και το σύστημα των ιδίων Πόρων. Ε, ο συνάδελφος Μπίγκε στην δική του αναλυτική έκθεση πρέπει να αναφερθεί και στο θέμα αυτό. Επίσης θα πρέπει οπωσδήποτε να εκφράσουμε και την άποψή μας ε, για το μελλοντικό μακροοικονομικό ε, σύστημα. Ε, γιατί η επόμενη δεκαετία θα είναι πάρα πολύ σημαντική. Κατά την άποψή μου έχει γίνει καλή πρόοδος τα τελευταία χρόνια ε, και έχουμε επιβάλει και κάποιες, ε, κάποια προαπαιτούμενα όσον αφορά τα μικροοικονομικά, χρηματοοικονομικά συστήματα και θα πρέπει ε, ε, οπωσδήποτε ας πούμε ε, να πούμε ότι εδώ έχουμε ένα ποσοστό της τάξης του 60 της όσον αφορά την επιχορήγηση που θα πρέπει να καταβάλλεται. Είμαι διατεθειμένος να συζητήσουμε το, το θέμα αυτό. Αναφερόμαστε στη μακροοικονομική συνδρομή. Ε, ε, και οπωσδήποτε ε, θα πρέπει οι, οι διαπραγματεύσεις να είναι πιο σοβαρές και πιο απαιτητικές έτσι ώστε το ρυθμιστικό πλαίσιο να είναι πιο συγκεκριμένο. Είναι γεγονός λοιπόν, μια και μιλάμε εδώ για χρήματα, ότι και ο χρόνος είναι χρήμα, γι' αυτό λοιπόν δεν χρειάζεται και εγώ να μιλήσω περισσότερο. Έχουμε εδώ μια νομοδότηση πολύ συγκεκριμένη. Σας ζητώ λοιπόν να δουλέψουμε όλοι μαζί για την γνωμοδότηση αυτή, ε, ε, να υπάρχουν, έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μια συνενετική ε, λύση, συμβιβαστικές τροπολογίες. Θα έχουμε δύο δυνατότητες ανταλλαγής απόψε... όσον αφορά το, την, τις τροπολογίες 27-28 Σεπτεμβρίου και βεβαίως περιμένω τις παρατηρήσεις σας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος. Και τώρα θα δώσω τον Α, λόγο. Περνάμε στους κοιοδες απο Από δύο-δυόμιση λεπτά ο καθένας. Ο κύριος Ρουιμπίκ είναι ο πρώτος. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ συνάδελφε Σόλτς. Ο επόμενος προϋπολογισμός νομίζω θα είναι ακόμα πιο δύσκολος από τον προηγούμενο που διαπραγματευτήκαμε. Έχουμε μια σκληρή ομάδα που επιμένει στο 1% και η συζήτηση για τους ιδίους πόρους είναι πολύ σημαντική. Μην το ξεχάσουμε αυτό. Και σίγουρα παίζουν και οι δασμοί μεγάλο ρόλο. Σε αυτό το τομέα τα έσοδα είναι 22 δις, περίπου 15% δηλαδή του συνολικού προϋπολογισμού και αυτό θα ενισχύσει τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Από το 17 στο 18 οι ήδη πόροι αυξήθηκαν κατά 6,41%. Οπότε έχουμε αυξημένα έσοδα αυτή τη στιγμή. Το πρόβλημα που τίθεται βέβαια είναι ότι οι φορολογικές απάτες πολλές φορές δεν αντιμετωπίζονται. Η ΟΛΑΦ μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ακολουθήσουν μια, θα εισαγάγουν, ε, άρχισαν ήδη δηλαδή κατά της Βρετανίας μια διαδικασία ε, φορολογικών παραβάσεων. Από το 12 μέχρι το 17, 2,7 δις ευρώ χάθηκαν ε, σε ό,τι αφορά τα φορολογικά έσοδα, κυρίως ε, λόγω των ε, λαθασμένων τιμολογίων και ε, λάθος ε, ε, δηλώσεων από την Κίνα και το λαθρεμπόριο τσιγάρων είναι μεγάλη ζημία και εκεί έχουμε μεγάλη απώλεια εσόδων. Γι' αυτό χαιρετίζω την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, το κόστος ε, ε, ερευνών από ε, να μειωθεί από το 20% στο 10% πράγμα που σημαίνει ότι ο νοσιακός προϋπολογισμός ε, μπορεί να ε, φτάσει στο 90% κάλυψη των εσόδων. Είναι σημαντικό ότι μπορέσαμε να βρούμε τρόπους για να αυξήσουμε τα έσοδα από τον ΦΠΑ ε, σε σχέση με το, το 17 είχαμε 16 δις και τώρα έχουμε αύξηση των ποσών από τον ΦΠΑ και έχουμε επίσης ε, και από τον ψηφιακό ε, τομέα δυνατότητες μεγαλύτερης ίσπραξης, πράγμα που διευκολύνει και τις ΜΜΕ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε σχέση με το σημείο 6, αυτό που ε, αναφέρεται στους αυξημένους πόρους για την πολυμέρεια και τις κανονιστικές ρυθμίσεις του παγκοσμίου εμπορίου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θα ενισχύσουμε και τις κοινοβουλευτικέ μας ε, δραστηριότητες σε σχέση με τον ΠΟΕ και πιστεύω ότι μαζί μπορούμε ε, να κάνουμε ορισμένες χρήσιμες αναφορές σε σχέση με τον πολιετές πλαίσιο. Αλέσια Μόσκα. Ευχαριστώ. τον εισηγητή για την καλή γνωμοδότηση. Συμμερίζομαι πολλές απόψεις που αναφέρονται στη γνωμοδότηση. Πρώτα απ' όλα ότι συμφωνούμε να διατηρηθεί η ευελιξία σε σχέση με το εξωτερικό δημοσιονομικό μέσο. Συμφωνούμε επίσης ότι μπορούμε να κινηθούμε μέσα στα πλαίσια ε, των ε, στόχων βιώσιμης ανάπτυξης, της αποφάσεις μας και τονίζω ε, ένα στοιχείο που ενδιαφέρει ιδιαίτερα να βελτιώσουμε τις αξιολογήσεις και εκ των προτέρων και ενδιάμεσων και εκ των υστέρων σε αυτό το πλαίσιο, λαμβάνοντας υπόψη το ε, ε, θεματολόγιό μας που είναι τόσο σημαντικό για μας. Επίσης, και τους ε, στόχους βέβαια ε, βιώσιμης ανάπτυξης. Επίσης, ε, ε, θα ωφεληθούμε από τις εταιρικέ σχέσεις ε, τις εμπορικές. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να προωθήσουμε το εμπόριο ε, μέσα από εκεί χρησιμοποιώντας όλα τα στοιχεία και τους πόρους που διαθέτουμε. Οι εσωτερικές συμβουλευτικές ομάδες είναι πάρα πολύ σημαντικό μέσον και χρήσιμο για να έχουμε ε, αποτελεσματική παρακολούθηση της διαδικασίας εφαρμογής υλοποίησης, αλλά ε, ε, ανησυχούμε διότι υπάρχει μία μείωση στους οικονομικούς, δημοσιονομικούς πόρους για το μέσον αυτό. Γι' αυτό ζητούμε αυξημένους πόρους και για το μέσον αυτό θα προτείνουμε νέα τροπολογία για το ε, Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, γιατί ε, ε, δεν είναι επαρκής η χρηματοδότηση, πιστεύομαι. Είναι μειωμένο ο υπολογισμός του. Επίσης, το ψηφιακό εμπόριο θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί επαρκώς για να υλοποιηθούν όλες οι σχετικές δράσεις που προβλέπονται στην απόφασή μας. Ε, εξωτερική δανειοδότηση θα παίξει μεγάλο ρόλο για να αντιμετωπίσει τους, τα αίτια της μετανάστευσης και χρειαζόμαστε πόρουσε για να αντιμετωπίσουμε τους ε, εκτοπισμένους. Πιστεύουμε λοιπόν ότι και εδώ θα πρέπει να ε, κάνουμε σχετικές τροπολογίες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Δυστυχώ οι άλλοι σκιώδεις δεν είναι παρόντες και δεν βλέπω να θέλει κανείς άλλο τον λόγο. Οπότε, κομισιόν παρακαλώ. Κυρία Σοφία Μουνιώθ. Αλβαράν, επικεφαλή πόρων και στρατηγικού σχεδιασμού της Γενική Διεύθυνση Εμπορίου της Trade. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τον εισηγητή, καθώς και τα μέλη της Επιτροπής για την υποστήριξη. Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια όσον αφορά τους κύριους στόχους της εμπορικής μας πολιτικής. Και εμείς, όπως εσείς, υποστηρίζουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό το μηχανισμό εταιρική σχέσης και τους άλλους μηχανισμούς, το προσχές ΠΔΠ, ήταν ένας από τους βασικούς μας στόχους στη διάρκεια της διαδικασίας κατάρτισης του επομένου ΠΔΠ, πολύ βασικό για την εμπορική πολιτική, γιατί είναι ένας από τους λίγους μηχανισμούς που μας επιτρέπουν να υπεραμεινόμεθα με τρόπο θα λέγει επιθετικό των ε, συμφερόντων της Ένωσης πέρα από τα εργαλεία αναπτυξιακής φύσης υπέρ της ε, βιώσιμης ανάπτυξης, την ισότητα των φύλων. Είναι τομείς όπου δεν μπορούμε αναγκαστικά να, να παράσουμε χρηματοδότηση μέσω των κλασικών μηχανισμών. Μπορούμε όμως να το κάνουμε εδώ και αυτό είναι ευτυχές. Τα συζητήσαμε αυτά για μακρόν με τι άλλε γενικέ διευθύνσει που έχουν σχέση με εξωτερικέ σχέσει και είπαμε ότι έτσι θα προχωρήσουμε. Ο μηχανισμό εξωτερική σχέση πρέπει να συνεχιστεί, να έχει το ίδιο ποσό, το ίδιο ύψος χρηματοδότηση για να χρηματοδοτήσουμε παρόμοιε δράσεις. Αυτά που κάναμε και τα περασμένα χρόνια. Έτσι θα μπορέσουμε λοιπόν να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε διάφορες χώρες στο πλαίσιο του προσεχούς ΠΔΠ. Συμφωνώ επίση ότι έχει σημασία η Γενική Διεύθυνση Trade και το εμπόριο γενικά να, έχει, να έχουν το δικό τους προϋπολογισμό, όπως έγινε και με το τρέχον ΠΔΠ. Έναν προϋπολογισμό τον οποίο θα διαχειρίζεται η Κομισιόν. Έναν προϋπολογισμό ο οποίος θα είναι εκτός του νέου εξωτερικού χρηματοδοτικού μέσου δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε τον ίδιο τρόπο με τα άλλα αναπτυξιακά εργαλεία. Αν το καταφέρουμε αυτό θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε διάφορες δράσεις όπως την αξιολόγηση που το τονίσετε κι εσείς, αξιολόγηση καθώς και καλύτερες σχέσεις, να έρθουμε πιο κοντά με τους εξωτερικούς μας εταίρους, τους πολίτες και αυτό είναι πολύ βασικό στην εξωτερική μας πολιτική και στην πολιτική για το εμπόριο και από εκεί πέρα βέβαια να υποστηρίξουμε διάφορους διεθνείς οργανισμούς στο πλαίσιο της βοήθειας για το εμπόριο, όπως λέμε. Αν γίνουν οι προτινόμενες μειώσεις, θα μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε το νέο μέσο. Οπότε, ευχαριστώ πολύ. Ε, νομίζω ότι συμπεριλάβατε στην έκθεση αυτά τα οποία υποστηρίζουμε και εμείς. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Επειδή έχουμε λίγο χρόνο, ε, να θέσω δύο ερωτήματα στην Κομισιόν. Πρώτον, γιατί ένα μόνο ταμείο για τις εξωτερικές σχέσεις. Είπατε ότι είστε πεπισμένοι ότι θα κάνουμε τα ίδια που κάναμε και στο παρελθόν. Όμως υπάρχει ένα πρόβλημα εδώ. διότι το μερίδιο των πόρων για το εμπόριο, οι σχετικές γραμμές δηλαδή στον υπερπολισμό, αν ε, τα συγκρίνουμε με τα αναπτυξιακά, ε, είναι πολύ περιορισμένα. Και υπάρχει ο φόβος ότι θα μείνουμε πίσω εμείς, η πτυχή εμπόριο δηλαδή. Δεύτερον, η σχέση εμπορικής πολιτικής Εσωτερικής πολιτική και το Ταμείο προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση. Θυμάστε την περίφημη ανακοίνωση της Κομισιόν όπου έλεγε ότι η παγκοσμιοποίηση έχει ωφέλη, ωφέλη αλλά ωφελήματα μάλλον και ε, προκλήσεις, δηλαδή προβλήματα, για να το πούμε με το όνομά τους, και ότι αυτά πρέπει κάπως να αντιμετωπιστούν. Αυτή είναι η εξωτερική διάσταση που αφορά την αναπτυξική βοήθεια, τις εμπορικές συμφωνίες κλπ. Αλλά υπάρχει και μια εσωτερική διάσταση. Την οποία μάλλον έχουμε παραγνωρίσει, θα λέω, υποτιμήσει. Έχετε κάποιες προτάσεις για να δούμε πώς θα ασχοληθούμε πιο σοβαρά με αυτή την εσωτερική διάσταση, πώς θα κάνουμε κάτι δηλαδή για τις επιπτώσεις στο εσωτερικό της ε, Ένωσης από την παγκοσμιοποίηση. Επίση, αυτό που είπε και ο κ. Ζουία, για την τελωνία, ποια είναι η θέση της Κομισιόν εν προκειμένου. Ιδιαίτερα εν ώψη του Brexit και της πρότασης της Βρετανικής κυβέρνησης να ισχύσουν δύο διαφορετικά μέτρα και σταθμά. Άλλα για το Ηνωμένο Βασίλειο, άλλα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποια είναι η άποψη τη Κομισιόν αυτού. Είναι ρεαλιστική αυτή η προοπτική. Και τέταρτον, τι γίνεται με το προσωπικό της γενική διεύθυνση Trade. Από ό,τι ξέρω, έχει επιβληθεί μια μείωση 2%. Αυτή αφορά και την Γενική Διεύθυνση Trade. Τώρα, όσον αφορά την αύξηση των διαπραγματεύσεων, έχουμε ένταση των διαπραγματεύσεων, έχουμε εμπορικέ διαφορές. Τι λέτε γι' αυτό. Θα καταφέρει το προσωπικό της ε, DigiTrade. Περισσότερο αντικείμενο, περισσότερη ύλη, λιγότερο προσωπικό. Κομισιόν, θα προσπαθήσω να απαντήσω στα ερωτήματα που θέσατε. Θα κάνω ό,τι μπορώ. Για το πρώτο, Πώ θα φροντίσουμε να διατηρήσουμε τον προπολογισμό μας στα ίδια επίπεδα. Δεν είμαστε 100% βέβαιοι. Ο κ. Σόλτς ανέφερε τα νέα στοιχεία του νέου μέσου. Ε, είπε ότι υπάρχει ευελιξία μέσα στα πλαίσια του ενιαίου μηχανισμού. Θα υπάρχει όντω ευελιξία, θα μπορούν να μεταφερθούν πόροι από το ένα αντικείμενο στο άλλο. Όμω, εν γέννη, θα έλεγα ότι οι στόχοι όσον αφορά το εμπόριο ως τώρα τουλάχιστον προστατεύθηκαν, έχουμε διάφορους μηχανισμούς στη διάθεσή μας όσον αφορά την εταιρική σχέση νομίζω πίνησα αλλά λίγο πολύ το ίδιο ποσό που χρησιμοποιήθηκε για τα του εμπορίου προέρχεται από τα αναπτυξιακά που αφορούν τις χώρες ΑΚΕ είτε αφορούν την εταιρική σχέση κλπ. Θέλω να πω δηλαδή ότι τα ίδια εργαλεία θα συνεχίσουν να υπάρχουν και να χρηματοδοτούνται βάσει των νέων προτάσεων, ούτω ή άλλω. Και όλα αυτά μαζί με τα αναπτυξιακά ταμεία. Είναι υπό την ομπρέλα των αναπτυξιακών εργαλείων ούτως ή άλλως. Τώρα, όσον αφορά τα νούμερα, τα πρώτα νούμερα που είδαμε, οι πρώτες ε, κατανομές, δείχνουν ότι υπάρχει αύξηση της χρηματοδότησης για το σύνολο των εργαλείων. Δεν είδαμε μείωση για τους προπολογισμού που μας αφορούν ως τώρα τουλάχιστον. Οπότε αυτά προς το παρόν, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Δεν έχουμε διαπιστώσει μειώσεις. Αντιθέτως, είδαμε αυξήσεις και σε κάποιες άλλες θέσεις απλώς διατηρείται ο ίδιος προπολογισμό, Ο στα ίδια επίπεδα. Δεύτερη ερώτηση παγκοσμιοποίηση και το σχετικό ταμείο. Η αξιολόγησή μας, η εκτίμηση της πρότασης για το ταμείο είναι ότι από εδώ και πέρα θα είναι ακόμη ευκολότερο με το νέο ταμείο να αντιμετωπίσουμε τις επιπτώσεις διαφόρων εμπορικών συμφωνιών στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για έναν μηχανισμό πιο ευέλικτο σε σχέση με αυτόν υπό το τρέχον πιδελταπή και αυτό για μας είναι θετική εξέλιξη. Θα δείξει όμως, θα δούμε πώς θα λειτουργήσει το πράγμα στην πράξη. Πάντως, στα χαρτιά τουλάχιστον όπως λέμε, φαίνεται ότι πρόκειται για ένα πιο ευέλικτο εργαλείο, το οποίο θα μας επιτρέψει να συνεχίσουμε ε, όχι μόνο να υποστηρίζουμε στα ίδια επίπεδα, αλλά και να εντείνουμε την υποστήριξή μας των προσπαθειών αντιμετώπιση των επιπτώσεων της παγκοσμιοποίησης. Ως υπηρεσία της Κομισιόν δεν μπορούμε παρά να συμφωνήσουμε. Να συμφωνήσουμε μαζί σας για την ανάγκη διερεύνηση της υπόθεσης από την Όλαφ. Τώρα η έρευνα αυτή, η διερεύνηση της υπόθεσης συνεχίζεται. Δεν έχει καταλήξει, θα δούμε ποιο θα είναι το τελικό αποτέλεσμα. Όμως, η συναδελφή της Όλαφ, όπως γνωρίζετε, συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις οι συμφωνίε περιλαμβάνουν διατάξει που προσπαθούν να προλάβουν την εμφάνιση προβλημάτων. Έχουμε διάφορα θέματα, τους κανόνες προέλευσης και καταγωγής. Είναι πράγματα τα οποία λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας στις εμπορικές συμφωνίες και τα, φροντίζουμε να είστε βέβαιοι σε όλες τις εμπορικές μας αν και δεν, ε, όπως καταλαβαίνετε, δεν πρόκειται για τις πιο εύκολες διατάξεις. Ούτε είναι εύκολο να τις διαπραγματευτείς. Και τέλος, όσον αφορά το προσωπικό της Γενικής Διεύθυνσης Trade και τι γίνεται με τον αυξανόμενο φόρτο εργασία, τι ε, διαπραγματεύσει για την εφαρμογή τη μιας ή τη άλλη συμφωνία κλπ. Κοιτάξτε, υπάρχει πίεση. Ε, υπάρχει έλλειψη προσωπικού εμείς ζητάμε εδώ και καιρό αύξηση των ανθρωπίνων πόρων. Το ζητήσαμε σε όλους τους τελευταίους ε, προϋπολογισμούς. Μας έκαναν μια μικρή αύξηση. Τώρα για φέτος ζητήσαμε τουλάχιστον να μην γίνουν περικοπές στο τέλος του έτους γιατί αυτό θα μας επηρεάσει σαφώς αρνητικά. Δηλαδή όχι μόνο δεν θα γίνει αύξηση αλλά θα περικοπεί και όλες το προσωπικό. Λοιπόν, υπάρχει πίεση όσον αφορά το προσωπικό, αλλά εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ελοπίσουμε τους στόχους μας. Θα συνεχίσουμε να ζητούμε πάντως ενίσχυση του προσωπικού τα προσεχή έτη, λόγω κυρίως της εφαρμογής των διαφόρων συμφωνιών ελευθερού εμπορίου που διαπραγματευόμεθα αυτή τη στιγμή. Εξαρτάται όμως από το πώς θα πάει η κατάσταση με τις ΗΠΑ θα δούμε αν θα καταφέρουμε να ενισχυθούμε με επιπλέον προσωπικό. Θα παρακολουθούμε την κατάσταση, εννοείται. Μέχρι στιγμής πάντως η Κομισιόν, όπως προείπα, μας έδωσε κάποια μικρή ενίσχυση του προσωπικού για να μπορέσουμε να τα καταφέρουμε να αντεπεξέλθουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, κύριος Προύστο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα ε, να αναφερθώ στο τελευταίο στοιχείο ε, το οποίο ανέφερε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δηλαδή την ενίσχυση ε, του προσωπικού της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίου, όπως πολύ συχνά έχω πει. Ε, είναι καλό να υπογράφονται συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου, αλλά ακόμα καλύτερο είναι να γίνονται σεβαστές οι συμφωνίες αυτές. Ε, η, η σημερινή περιπλοκότητα και πολυμέρεια, και το είπατε κι εσείς, ε, συμπεριλαμβάνονται όλο και περισσότερες ρήτρε στις εμπορικές συμφωνίες. Και επομένως, όταν δει κανεί τον αριθμό των μελλοντικών αυριανών, μεθαυριανών, ας πούμε, συμφωνιών που ελπίζω ότι θα υπογραφούν, αναρωτιέμαι πώς με σταθερούς ανθρώπινους ε, πόρους ε, μπορούμε να είμαστε αποτελεσματική ακόμα και στις διαπραγματεύσεις γιατί ε, θυμάμαι όταν ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις TTIP ε, ήταν πολύ λιγότερη ε, πολύ ε, λιγότερο αριθμητικά η αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής δηλαδή πλευράς από την Αμερικανική Εμβάση. περιπτώσει κυρίως ο έλεγχος πώς θα γίνεται γιατί με αυτόν τον τρόπο αποδεικνύουν την, την αποτελεσματικότητά τους οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και επομένως θα πρέπει πολύ σοβαρά να δούμε το βάρος το οποίο έχει το προσωπικό της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίου. Θέλετε να πείτε κάτι? Ίσως, ίσως να κάνω μία μικρή παρατήρηση, λέει εκπρόσωπος της Κομισιόν. Η υλοποίηση της ε, συμφωνίας δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου. Ε, ε, είναι ένα ευρύτερο πλαίσιο. Βεβαίως έχουμε και επιτόπου, έχουμε και στην έδρα μας προσωπικό που εργάζεται, έχουμε όμως και επιτόπου και έχουμε επίσης και προσωπικό που προέρχεται από άλλες γενικές διευθύνσεις που εμπλέκεται άμεσα ή έμεσα στις ε, συμφωνίες και τις διαπραγματεύσεις. Είναι γεγονός ότι πρόκειται για θέματα ε, σοβαρά ε, που παίρνουν χρόνο, αλλά να σας πω ότι όσον αφορά ας πούμε, το τμήμα της ανάλυσης που είναι και το πιο χρονοβόρο, πολύ συχνά μοιραζόμαστε το βάρος με άλλα μέσα ε, Επίσης, μέσω εταιρικών σχέσεων ε, έχουμε χρηματοδοτήσει ε, δομές οι οποίες μπορούν να υποστηρίξουν οικονομικά την εφαρμογή, υλοποίηση των ε, συμφωνιών μας και με μια καλή διαχείριση των πόρων θα μπορέσουμε να διαχειριστούμε καλά και τις υφιστάμενες εμπορικές συμφωνίες αλλά ευελπιστούμε και τις μελλοντικές. Ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ λέει ο, ο Πρόεδρος. Ε, ναι, αλλά φαίνεται ότι από πλευρά ε, των ΗΠΑ δεν χρειάζονται και πολλοί για να ολοκληρώσουν εμπορική συμφωνία. Ένα και καλό αρκεί. Ελπίζω αυτό να μην γίνει ο κανόνα όμω. Ευχαριστώ την Κομισιόν για τι πρόσθετες πληροφορίε και την ανταλλαγή απόψεων που είχαμε. Είναι σύνθετες οι προκλήσεις στο νέο δημοσιονο... πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και έχουμε μια νέα ε, προσέγγιση ώστε να συμπεριλάβει όλα τα στοιχεία. Αυτό για τον νομοθέτη ε, θέτει και θέμα ελέγχου, θέμα άσκησης επιρροής στα μέσα αυτά και το πώς κατανέμονται τα κονδύλια Πρέπει να υπάρχει διαφάνεια και το Κοινοβούλιο χρειάζεται να παρακολουθεί τι γίνεται όταν εφαρμόζονται οι εμπορικές συμφωνίες. Δεν μίλησα και για το ξέπλυμα χρήματος. Θα πρέπει οι εμπορικές συμφωνίες να είναι τόσο ακριβείς ώστε να μην ε, χρησιμεύουν για να γίνουν παράτυπα είσοδοι στην αγορά. Όλα αυτά πρέπει να τα δούμε. Χρειάζεται μεγαλύτερη ακρίβεια και επίσης και το Κοινοβούλιο θα πρέπει να έχει σωστή οριζόντια συνεργασία με τις άλλες επιτροπές όταν υπάρχει ένα τέτοιο μέσον και χρειάζεται μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση των συναδέλφων που πρέπει να γνωρίζουν ότι η εξωτερική μας εμπορική πολιτική σχετίζεται με πολλά άλλα θέματα που αφορούν το εσωτερικό της Ένωσης. Ε, μαζί με την Επιτροπή Προϋπολογισμού συμφωνήσαμε να συναντηθούν οι σκιώδεις ε, υπεύθυνοι για διάφορα θέματα, ούτως ώστε να ενημερώσουν επαρκώς το Κοινοβούλιο σχετικά με το τι, πώς θα αντιμετωπίσουμε το πολιετές πλαίσιο ε, την επόμενη δεκαετία. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για την εμπιστοσύνη των πολιτών. Είναι σημαντικό αυτό. Αυτό σε τελευταία ανάλυση μετράει. Αν μας εμπιστεύονται, ε, προσβλέπουμε επικοδομητική συνεργασία, επικοδομητική συνεργασία με τους σκιώδεις και ελπίζουμε ότι η γνωμοδότησή μας θα μπορέσει να συμβάλλει σημαντικά στις μελλοντικέ συζητήσεις στο Κοινοβούλιο. Ε, περιμένω στενότερη ακόμα συνεργασία. Ε, θα έχουμε νομίζω στις 27 Σεπτεμβρίου μια ακόμη ανταλλαγή απόψεων. Ευχαριστώ. Η προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών είναι η 7η ε, Σεπτεμβρίου στις 12 το μεσημέρι. Ωραία. Και πάω στο επόμενο σημείο, το 21, στην ημερήσια διάταξη. Πρόκειται για την ετήσια έκθεση για τους φραγμούς στο εμπόριο και τις επενδύσεις. Υπάρχει εδώ μια αβεβαιότητα. Η έκθεση είναι σημαντική. και τα αποτελέσματα της έκθεσης ε, συνιστούν προκλήσεις σε πολλούς τομείς του εμπορίου και των επενδύσεων. Και με ενδιαφέρον θα ακούσουμε τις λεπτομέρειες της έκθεσης. Ο κύριος Φρανσίσκο Περές Κανάντο, ε, προϊστάμενος μονάδας, θα κάνει την παρουσίαση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, χαίρομαι που είμαι εδώ για να παρουσιάσω τα βασικά στοιχεία της φετινής έκθεσης που είναι, η, περιλαμβάνει τις προσπάθειες της Ένωσης να καταρρύψει τους φραγμούς. Η... Πρέπει στην αρχή να θυμίσω με κάποια πράγματα που είναι πολύ σημαντικά πιστεύουμε, βασικά μηνύματα για φέτος δηλαδή. Πρώτον, αντιμετωπίζουμε περισσότερους φραγμούς από ποτέ. Ε, αύξηση προστατευτισμού. Δεύτερον, αυξάνει ο προστατευτισμός, αυξάνουν και οι προσπάθειές μας όμως. Απαλείψαμε περισσότερους φραγμούς από οποτεδήποτε στο παρελθόν και έχουμε ρεκόρ ε, πάνω από 4,8 δις το χρόνο ε, αύξηση είχαμε και αυτό επηρεάζει πολλούς, κυρίως τις ΜΜΕ και αυτό αποδεικνύει και την αυξανόμενη δέσμευσή μας υπέρ μια στρατηγικής ε, ανταγωνισμού, θέσεων εργασίας κλπ. Έχουμε τη στρατηγική για την πρόσβαση στην αγορά, αναθεωρήσαμε τον τρόπο λειτουργίας μας για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις. Παράλληλα με αυτό το μήνυμα έχω και κάποιες κακές ειδήσει. Δηλαδή, στο μέλλον θα αντιμετωπίσουμε οπωσδήποτε μια περίοδο μεγάλων προκλήσεων και πρέπει να διπλασιάσουμε τις προσπάθειες να αξιοποιήσουμε στο μέγιστο αυτή τη στρατηγική για την πρόσβαση στην αγορά γιατί βλέπουμε ε, ότι αυξάνεται ο προστατευτισμός. Τώρα, σε αυτές τις βελτιωμένες ε, προσπάθειες ε, ε, μπορεί να παίξει και το Κοινοβούλιο σημαντικό ρόλο. Να θυμίσω κάτι σε όσους δεν γνωρίζουν πολύ καλά αυτές τις εργασίες, πώς δηλαδή λειτουργεί η, πρόσβαση στην, η στρατηγική για την πρόσβαση στην αγορά. Οι εταιρείε ε, ε, έρχονται στην Κομισιόν, εντοπίζουν τους φραγμούς που εμποδίζουν την είσοδό του στην αγορά όπως πιστεύουν και μετά έχουμε στοχοθετημένα μέτρα ε, εξατομικευμένα και εδώ και στις αντιπροσωπείες που χαράζουν την απαραίτητη στρατηγική, lobbying, διπλωματικές προσπάθειες και πολλά άλλα. Χάρη σε αυτή την κοινή δουλειά με τις επιχειρήσεις φέτος είδαμε ότι σαφώς αυξάνεται ο προστατευτισμός, έχουμε ρεκόρ 67 νέων εμποδίων, ε, οπότε έχουμε συνολικά 396 εμπόδια ε, που είναι πολύ μεγάλος αριθμός και επηρεάζει ε, σε τάξη μεγέθους διψήφιο δισεκατομμυρίων. Τώρα, η Κίνα έχει τη μεγαλύτερη αύξηση των εμποδίων τον, ε, το 2017, ακολουθείται από την Ρωσία, Νότια Αφρική, Ινδία και Τουρκία. Και η μεσογειακή περιοχή ε, επίσης προστίθεται που αύξησε τα εμπόδια για τις επιχειρήσεις μας. Τώρα, σε επίπεδο τομεακό, ε, διατροφικός τομέας γεωργικά προϊόντα, ε, αντιμετωπίζει μεγάλα εμπόδια, ε, τα, τα δέρματα, τα χημικά, ε, ηλεκτρονικά, τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας. Ε, εμείς, ε, επειδή θυγόμεθα, αυξήσαμε τις προσπάθειες και ε, ανταποκριθήκαμε στη δέσμευσή μας. Είχαμε 40 πέντε νέους, ε, νέα εμπόδια τα οποία τα καταργήσαμε, διπλάσιος αριθμός από ό,τι πέρσι και έτσι οι καταργηθέντες ε, φραγμοί είναι 88, αριθμός ρεκόρ επίσης. Αυτό ε, δεν επηρέασε ένα συγκεκριμένο τομέα, αλλά κάλυψε πολλούς περισσότερους τομείς. Αυτό απέδειξε ότι η στρατηγική μας ε, λειτουργεί και για τον ε, τομέα των, ε, ε της αεροναυπηγικής και, κεραμικών πλακιδίων κλπ. Από τα μεγάλα μέχρι τα μικρά πρόσθετες εξαγωγές που κερδίσαμε χάρη στις προσπάθειές μας. Τουλάχιστον 4,8 δις πρόσθετες εξαγωγές. Βέβαια τα νούμερα δεν σημαίνουν τίποτα, πρέπει να τα βάλουμε μέσα σε ένα πλαίσιο. Σας λέω λοιπόν ότι αυτό είναι ένα, δύο ή τρία, ανάλογα με τη χώρα που θα πάρουμε, του, ε, παραπάνω από το εμπόριο που πραγματοποιείται μέσα από τη ΣΕΣ. Οι, ΣΕΣ ε, είναι, ε, αποφέρουν έσοδα, αλλά υπάρχουν και πρόσθετα ωφέλη. Οι λύσεις που βρήκαμε για να λύσουμε τα προβλήματα ε, ωφέλησαν συγκεκριμένες επιχειρήσεις. Θέλαμε να δώσουμε ένα ανθρώπινο πρόσωπο σε αυτά τα ανοίγματα στην αγορά. Εδώ εξετάζω, τώρα εξετάζουμε πορτογαλική, μια ε, πορτογαλική εταιρεία που τη βοηθήσαμε να λύσει ένα πρόβλημα με την Τουρκία στον τομέα του χαρτιού ε, το, και υποστηρίξαμε ε, τις θέσεις εργασίας αυτής της επιχείρησης. Περίπου 900. Πώς έχουμε καταγράψει αυτές τις επιτυχίες. Πρώτον, ε, Είχαμε καλύτερο συντονισμό μεταξύ κομισιών, κρατών μελών, επιχειρήσεων που είναι πολύ σημαντικό. Χαράσε τη σωστή στρατηγική και ακολουθείται, καλύτερη ιεράρχηση των φραγμών, γιατί δεν μπορούμε ταυτόχρονα να ασχοληθούμε με όλους τους φραγμούς, επικεντρωθήκαμε στους σημαντικότερους και βελτιώσαμε την επικοινωνία και την ευαισθητοποίηση. Αυτές είναι ακριβώς οι μελέτες είναι, αυτό είναι το αντικείμενο της μελέτης που είχε ανατεθεί και ε, ευθυγραμμιζόμαστε προς τις προτάσεις της. Δύο ακόμα πράγματα να σας πω. Πρώτον, για να σας δώσω και ένα παράδειγμα, πρέπει να ξέρουμε και πρέπει να ε, φτάσουμε στις ε, ΜΜΕ. Γιατί πολλές φορές δεν ξέρουν τις δυνατότητες που έχουν για την πρόσβαση στην αγορά μέσα από τη στρατηγική μας. Είχαμε λοιπόν τις ημέρες πρόσβασης της αγοράς MAD είναι το ακρονίμιο, μην το χρησιμοποιείτε. Ε, είναι λοιπόν μια σειρά επισκέψεων που κάνουμε επί τόπου, όχι στις ε, ε, πρωτεύουσε, αλλά στις περιοχές, στις περιφέρειες που θίγονται από συγκεκριμένα προβλήματα και εκεί έχουμε επαφή με τις ΜΜΕ για να τους εξηγήσουμε τι πρέπει να κάνουν για να βοηθηθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με την πρόσβαση στην αγορά, στη Δανία, στην Ισπανία το κάναμε φέτος, θα πάμε στο τέλος του χρόνου στην Ολλανδία και κάθε χρόνο πάμε σε τρεις-τέσσερις χώρες ώστε να καλύψουμε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είπα στην αρχή ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να βοηθήσει. Πού θα πρέπει να διπλασιάσουμε τις προσπάθειες. Πρέπει να το κάνουμε. Γι' αυτό πρέπει να μας βοηθήσετε. Πώς θα μας βοηθήσετε, σημαντικά μάλιστα, για να καταρρύψουμε τα εμπόδια στην αγορά, στην πρόσβαση στην αγορά. Να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση, η ενημέρωση. Εσείς έχετε επαφή με τις εκλογικέ περιφέρειες, με τους εκλογείς σας ενημερώστε για την εταιρική σχέση για την πρόσβαση στην αγορά που βοηθάει και έχουμε ε, υπηρεσίες που βοηθούν χιλιάδες επιχειρήσεις κάθε χρόνο να τους φέρετε σε εμά αν είναι δυνατόν. Επίσης παίζεται πολύ σημαντικό διπλωματικό ρόλο το, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εσείς που ταξιδεύετε στο εξωτερικό, ε, μπορεί να ασκήσει τεράστια επιρροή στους εταίρους. Μεταφέρετε τα μηνύματα όταν πάτε στην Κίνα, όταν πάτε στις Ηνωμένες Πολιτείες, όταν πάτε στην Τουρκία, να ενημερώσετε τα ε, θέματα αυτά είναι βασική προτεραιότητα, κορυφαία. Η πρόσβαση στην αγορά για τις επιχειρήσεις μας, για την ανάπτυξη, την οικονομική μεγέθυνση, την ανταγωνιστικότητα. Δεν θέλω να σας φορτώσω με δουλειά, αλλά όταν ε, ήμουν επικεφαλής της αντιπροσωπείας ε, για εμπορικά θέματα, είχα εντοπίσει όλες αυτές τις ανάγκες. Τώρα ε, χρειάζονται τεράστιες προσπάθειες για να αντιμετωπίσουμε πιο δύσκολες καταστάσεις. Ε, οι επιχειρήσεις πρέπει να είναι βέβαιες ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Κομισιόν είναι στο πλευρό τους και ε, θα εργαζόμεθα για να καταρρύπτουμε εμπόδια καθόν χρόνων οι άλλοι τα δημιουργούν. Ευχαριστώ. Πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Δύο ερωτήσει. Βρίσκω πολύ ενδιαφέροντα τα όσα κάνετε για τις μικρομεσαίες. Το πραγματικό πρόβλημα φαίνεται να είναι αυτό. Δηλαδή, αυτό που κάνει η Κομισιόν και οι άλλοι ευρωπαϊκοί θεσμοί να ωφελήσουν τις μικρομεσαίες. Αυτό είναι και πολιτικό πρόβλημα, γιατί πολλοί δεν γνωρίζουν ποια είναι τα ωφελήματα από τα όσα έχει κάνει η Κομισιόν και η Ευρώπη γενικότερα. Πέρα από τις ε, ημέρες πρόσβεσης στην αγορά που διοργανώνονται υπάρχουν άλλοι μηχανισμοί, άλλα εργαλεία τα οποία θα μπορούσατε να αξιοποιήσετε. Δηλαδή, ο καθένας έχει τον ρόλο του, την ευθύνη του για να διαδώσει το μήνυμα και τις σχετικές πληροφορίες. Όμως, χρειαζόμαστε περισσότερα. Δεν νομίζω ότι αυτέ οι ημέρε πρόσβαση στην αγορά είναι αρκετέ για να καλύψουν όλε τι περιοχέ, για παράδειγμα. Να πάρω τη χώρα μου. Είναι τόσοι κλάδοι, τόσοι οι τομεί που είναι πολύ δύσκολο να του καλύψουμε όλου μόνο με αυτέ τι ημερίδε πρόσβαση στην αγορά. Η ερώτηση μου λοιπόν είναι, προβλέπετε κάτι άλλο, κάποια άλλα εργαλεία, επιπλέον εργαλεία. Δεύτερον, από νομοθετική απόψεως. Αυτό που κάνουμε εδώ. Και σχετικά με δύο συγκεκριμένου φακέλου. Η αξιολόγηση των επενδύσεων και ο μηχανισμό δημοσίων συμβάσεων. Τι σχέση έχουν αυτά με αυτό που κάνετε εσείς αυτή τη στιγμή σε διεθνές επίπεδο στην προσπάθειά σας να ανοίξετε νέες αγορές. Συγχαρητήρια και από μένα για τη δουλειά σας. Πολύ καλή έκθεση. Ε, και εγώ έχω ερωτήσει. Πρώτον, είναι αλήθεια ότι οι αντιπροσωπείε τη Επιτροπή σε τρίτε χώρε. Είμαι σίγουρο ότι κάνουν πολύ καλά. Ε, καλή δουλειά, αλλά θα μπορούσαν να βοηθήσουν περισσότερο. Και να βοηθήσουν και τι μικρομεσαίε στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, κυρίω με τα δασμολογικά θέματα. Και άλλη μια ερώτηση πιο συγκεκριμένη. Πιστεύετε ότι οι γενικέ διευθύνσει διαθέτουν τα απαραίτητα μέσα για να υποστηρίξουν τις επιχειρήσεις μας όταν βγαίνουν σε αγορέ τρίτων χωρών. Έχω μια ανησυχία εδώ με αυτά που βλέπω. Τι γίνεται λοιπόν με τα μέσα που τελικώς θα εξασφαλίσουν καλύτερη πρόσβαση στις αγορέ. Το λέω γιατί ξέρω ότι σε πολλές περιπτώσεις οι αντιπροσωπείε δεν έχουν τα μέσα για να αντιπεξέλθουν. Γι' αυτό και θέτω το ερώτημα. Μπορούμε να βελτιώσουμε τα μέσα, να αυξήσουμε τον προπολογισμό και πώς θα μπορούσαμε γενικότερα να βελτιώσουμε τη στρατηγική μας. Και κάτι άλλο, η πρόσβαση στην πληροφορία είναι πολύ σημαντική. Η Γενική Διεύθυνση Trade έχει κάνει πολλά. Εν τούτης, θεωρώ ότι υπάρχει ακόμη και σήμερα άγνοια σε πολύ μεγάλη κλίμακα μεταξύ των επιχειρήσεων για τους διαθέσιμους μηχανισμούς. Οπότε, Νομίζω ότι χρειαζόμαστε καλύτερο συντονισμό με τα κράτη-μέλη, με τι αντιπροσωπεί τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Χρειαζόμαστε περισσότερη συνεργασία για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την κατάσταση, να αξιοποιήσουμε καλύτερα τι προσπαθίε μα. Ε, Αλλιώ θα δούμε αυτά που είδαμε και φέτο. Ευχαριστώ. Πρόεδρος. Αναφέρεται, έχω και εγώ ένα ερώτημα, 67 νέα εμπόδια και άρση 45 αν δεν κάνω λάθος. Άρα συν 22 νέα εμπόδια είναι ο τελικός λογαριασμός. Είναι αυτό αντιπροσωπευτικό σε παγκόσμιο επίπεδο. Και κάτι παρόμοιο. Τα εμπόδια τι ρόλο και πώς συσχετίζονται με τη νέα κυβέρνηση στις ΗΠΑ. Συνδέεται και με τις προσπάθειες άλλων τρίτων χωρών να εισαγάγουν εμπόδια. Και κάτι για την Κίνα επίσης. Έχουμε θετικά παραδείγματα από το πρόσφατο παρελθόν, αλλά θέματα παραμένουν ανοιχτά προ συζήτηση. Ποια είναι η γενικότερη εκτίμησή σα όσον αφορά την Κίνα, Τη βλέπετε να ανοίγει, να είναι πρόθυμη να καθίσει σε διάλογο. Από στρατηγική απόψεω, πού πηγαίνει η Κίνα όσον αφορά τα εμπόδια. Κομισιόν. Σας ευχαριστώ πολύ για όλες αυτές τις ερωτήσεις. Οφείλω να συμφωνήσω με πολλά από τα όσα ακούστηκαν προηγουμένως. Η ε, κυρία Μόσκα προηγουμένως, ε, θα σας πω κάτι. Ρωτήσαμε τα κράτη-μέλη. Το 28. Ποιος ενδιαφέρεται να προχωρήσουμε αναπεριφέρεια, να πάμε σε όλες τις περιφέρειες, τα κράτη-μέλη και να εξηγήσουμε τι ακριβώς σημαίνει αυτό. Μην το πείτε πουθενά, αλλά η Ιταλία δεν ζήτησε να είναι στις προτεραιότητες. Και ας μείνει μεταξύ μας μυστικό. Αυτό σας δείχνει νομίζω και λίγο τους περιορισμούς ε, τους οποίους αντιμετωπίζουμε. Θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν αυτές ε, οι εκδηλώσεις ή αυτά τα, ε, στοιχεία ας πούμε ως πολλαπλασιαστές του αποτελέσματος. Θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι οι περιφερειακές οργανώσεις καθώς επίσης και τα επιμελητήρια τα οποία έχουν δυνατότητα προσέγγισης και ευαισθητοποίησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων να εμπλακούν. Θέλουμε διαρκή ε, επαφή ε, έτσι ώστε να προωθηθεί και ε, το, το μήνυμα. Θέλουμε όσλο και περισσότεροι από αυτούς τους ανθρώπους ε, να εμπλέκονται, να συνδέονται με το λογαριασμό μας, να ενημερώνονται. Είναι μικρά πράγματα. Η πρόσβαση αγοράς market access δεν αποτελείται, αν θέλετε, δεν σημαίνει κάτι το τεράστιο, το μεγάλο, αλλά σημαίνει τα μικρά αυτά πράγματα. και χρειάζεται χρόνος έτσι ώστε να ε, προσεγγίσουμε όλο και περισσότερες ε, επιχειρήσεις. Επίσης ενημερώνουμε ε, και μέσα από περισσότερες πληροφορίες από την ιστοσελίδα μας, από τη βάση μας στις Βρυξέλλες. Υπάρχουν πολλά εργαλεία, αλλά σας το λέω και το επαναλαμβάνω οπωσδήποτε, είναι μια διαδικασία που παίρνει χρόνο. Ε, η κυρία Γκαρθία Πινιέιρο ε, αναφέρθηκε στις εταιρικέ σχέσεις με τις ε, χώρες. Είχαμε μια καλή εμπειρία με την Ισπανία πριν από το καλοκαίρι μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρουσα η ερώτηση κυρία Μόσκα, αυτή που κάνατε, πώς δουλεύετε με φακέλους που είναι, πώς να τους πούμε, αμυντικοί φάκελοι ε, εγώ θα πρέπει να σας παραπέμψω στην εμπειρία που είχα στην Κίνα με την προηγούμενη δουλειά μας. Δουλειά μου. Είχαμε πολλές δυσκολίες ε, και όσον αφορά τις επενδύσεις και όσον αφορά τις δημόσιες ε, προμήθειες στην Κίνα. Σε πολύ υψηλό επίπεδο έβλεπαν ότι συζητούνται τα θέματα αυτά και η πρώτη πολιτική ερώτηση είναι πού βρίσκεστε, πού έχετε φτάσει όσον αφορά την, το investment screen και όσον αφορά και και τις δημόσιες προμήθειες. Ε, θα πρέπει οπωσδήποτε και ο δημόσιος τομέας να μας βοηθήσει να κάνουμε τη δουλειά μας και επομένως εγώ σας ζητώ να μας βοηθήσετε κατά την έννοια αυτή. Ξέρω ότι τα θέματα αυτά είναι δύσκολα αλλά παρόλα αυτά πρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, να ε, βοηθήσει γιατί ακριβώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παίζει εξαιρετικά μεγάλο ρόλο στην όλη διαδικασία. Η κυρία Ροδόγης Πινιέιρο τώρα ρώτησε κάποια πράγματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ερωτήσεις. Θα σας δώσω κάποια ε, παραδείγματα. Πάλι θα μιλήσω για την εμπειρία μου στην Κίνα και την αντιπροσωπεία εκεί πρέπει να πω ότι έχουμε την τύχη ε, να έχουμε ε, αρκετούς συναδέλφους ε, που ασχολούνται με τα θέματα αυτά. Έχουμε επίσης ένα κέντρο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και που αποκλειστικά στόχο και σκοπό έχει την βοήθεια, να δώσει βοήθεια στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις έτσι ώστε να επιτύχουν πρόσβαση στην αγορά. Δεν τα λύνει όλα, αλλά είναι ένα καλό παράδειγμα. Ε, και όσον αφορά την ε, Market Access Partnership που εξηγούσα προηγουμένως, ε, για κάθε κεντρικό πρόβλημα πρόσβασης αγοράς έχουμε εταιρική σχέση με εταιρείε επιτόπου που ενδιαφέρονται για το θέμα με την πρεσβεία των, των, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τους συναδέλφους που δουλεύουν επιτόπου, έτσι ώστε να δούμε όλοι μαζί με ποιο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο δηλαδή, μπορούμε να λύσουμε αυτό το πρόβλημα πρόβλημα πρόσβαση αγορά. Και κάνατε και μια δεύτερη ερώτηση, η οποία εν μέρει απαντήθηκε ήδη. Μιλάμε εδώ για εταιρική σχέση. Πρέπει να έχουμε στενή συνεργασία ε, ανάμεσα στους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έτσι ώστε πραγματικά να μπορέσουμε να ε, έρουμε τόσο τα μεμονωμένα εμπόδια φραγμούς. Ε, τώρα εσείς κύριε Πρόεδρε κάνετε ερωτήσεις οι οποίες χρειάζονται έτσι ε, πολύ σοβαρές ε, απαντήσεις, ανυψώνετε πάντα το επίπεδο. Ε, ε, εδώ οι εξελίξεις που αναφέρουμε ε, είναι του 17, είναι πριν από τις εξελίξεις που έλαβαν χώρα το, στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά καταδεικνύει παρόλα αυτά ότι κάποια από τα προβλήματα προσβασιμότητας και κάποια, κάποιοι από τους φραγμούς, ας πούμε, με την Κίνα έδειχναν ήδη την τάση που οδήγησε στα όσα συμβαίνουν τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και, εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά δείχνουν ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε σε οριζόντια ε, βάση ορισμένα προβλήματα εάν πράγματι θέλουμε να σταθεροποιηθεί εκ νέου ε, ο εμπορικός κόσμος. Και ε, ε, γι' αυτό λοιπόν εμείς θέλουμε οπωσδήποτε να δούμε την, τον εξυγχρονισμό του ΠΟΕ. Πρέπει οι κανόνες να είναι τέτοιοι έτσι ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις νέες καταστάσεις. Όσον αφορά νέες τάσεις σχετικά με αύξηση φραγμών περισσότερο από άλλους, δεν έχω συγκεκριμένους αριθμούς για φέτος, αλλά ε, μάλλον η απάντηση θα είναι θετική, δηλαδή υπάρχει ένα αποτέλεσμα ντόμινο ε, και είναι πολύ πιθανό να έχουμε πραγματικά αύξηση των φραγμών. Επίσης, ε, να πω ότι η Κίνα έχει μέχρι ένα μεγάλο μέρος κρατάει το κλειδί της λύσης του προβλήματος. Όπως ξέρετε, εμείς θέλουμε να υποστηρίξουμε την Κίνα στις μεταρρυθμίσεις και το άνοιγμα, αλλά παρόλα αυτά ξέρουμε ότι αυτές ε, οι κινήσεις για το άνοιγμα της αγοράς δεν έχουν γίνει ακόμα. Οι επιχειρήσεις μας τις, περισε... Ε, τις ε, περιμένουν ακόμα. Ε, ε, χρειαζόμαστε λοιπόν και ε, οπωσδήποτε μια στενετική θέση απέναντι στην Κίνα, αλλά και σταθερότητα όσον αφορά τις απαιτήσει και των δικών μας επιχειρήσεων. Είχαμε συνάντηση τον Ιούλιο με την Κίνα, στοιχεία πρόσβασης αγοράς για πρώτη φορά αναφέρονται ως ε, κύρια προτεραιότητα ε, στο ανακοινοθέν που ακολούθησε αυτήν την ε, συζήτηση, αυτήν την συνάντηση. Θα μου πείτε λόγια, είναι γραμμένα σε ένα χαρτί, αλλά παρόλα αυτά καταδεικνύει αυτή η πρώτη αναφορά ότι αναγνωρίζει και εκείνο ότι υπάρχει ένα ζήτημα. Βέβαια, πολλή δουλειά ακόμα μας περιμένει, πολλή δουλειά έχουμε ακόμα μπροστά μας. Ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Τελειώσαμε το 21. Σας έχω το σημείο στην ημερήσια διάταξη. Ευχαριστώ πολύ και προχωρούμε στο σημείο 22. Είχαμε μία αντιπροσωπεία του Χόκ στην Μπαγκόκ, στην, της Ταϊλάνδης, ε, μεταξύ 17 και 19 Ιουλίου του 18. Ήταν διαρευνητική αποστολή Καθυστερήσαμε τις εμπορικές μας διαπραγματεύσεις με την Ταϊλάνδη, όπως γνωρίζετε, λόγω των πολιτικών εξελίξεων και είχαμε και κάποια θέματα ε, με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είχαμε και από τη Σχετική Επιτροπή εκπρόσωπο και είχαμε ένα κοινό πρόγραμμα ε, για, για μία μέρα από τις τρεις. Ο μόνιμος ε, εισηγητή για την Ταϊλάνδη, ο κ. Προύστα, θα μα ενημερώσει. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Όπως είπατε και προηγουμένως, κάναμε την αποστολή αυτή 17 με 19 Ιουλίου. Εγώ ήμουν εκεί ως μόνιμος εισηγητής για την Ταϊλάνδη. Κάναμε δέα, όπως είπατε, και ad hoc παράλληλη ε, ε, αποστολή ε, με την Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου έτσι ώστε να δουν πώς έχει η κατάσταση με τα δικαιώματα του ανθρώπου. Θέλαμε να δούμε πώς έχει η οικονομική κατάσταση και πώς μπορούμε να βελτιώσουμε το μέλλον των εμπορικών μας οικονομικών σχέσεων με τη χώρα αυτή. Είχαμε σειρά συναντήσεων και θα ήθελα πραγματικά να συγχαρώ την Γραμματεία της Επιτροπής για τον τρόπο με τον οποίο ε, οργάνωσε αυτό το τόσο βαρύ αλλά τόσο ενδιαφέρον πρόγραμμα. Ε, ήρθαμε σε επαφή και με επιμελητήρια, ε, με ε, υπευθύνους επενδύσεων, κάποια Υπουργεία, Υπουργείο Εργασίας και Υπουργείο Εμπορίου και βεβαίως ήρθαμε σε επαφή με το σύνολο των πολιτικών μας εκπροσώπων επιτόπου και φυσικά με την πρεσβεία των, της Ευρωπαϊκής Δουλέψαμε εν παραλίλω, αλλά δεν θα αναφερθώ εγώ στα ανθρώπινα δικαιώματα, έστω και ε, σε όλες ε, τις ε, συναντήσεις εκφράστηκε κάποια ανησυχία, προβληματισμός όσον αφορά την αντιμετώπιση της Ταϊλάνδης για την οποία εφηρμόζονται αρχές και μέτρα που δεν εφαρμόζονται σε άλλες χώρες με τις οποίες έχουμε επαφές και μάλιστα συνάπτουμε και εμπορικές συμφωνίες. Το χρονοδιάγραμμα ήταν σημαντικό και μπλοκάρισε κατά κάποιο τρόπο και την ε, συνέχεια των, ε, συνέχιση ε, των εμπορικών διαπραγματεύσεων. Μου είπαν ότι μετά από την στέψη του βασιλέως θα μπορούσαν να συνεχίσουν οι διαπραγματεύσεις, αλλά στο πρώτο εξάμεινο του 19 θα γίνουν και εκλογές στην Ταϊλάνδη. Σε γενικές γραμμές, μέχρι το τέλος του έτους η Ταϊλάνδη θα αναλάβει την Προεδρία της ΕΝΑΣ και επομένως θα όπως μας είπαν και όλοι οι οικονομικοί ε, πρωταγωνιστές, ε, θα γίνει ε, κεντρικό στοιχείο της Ασίας. Έχει πολύ καλή θέση μετά από την Κίνα και την Ιαπωνία και την Κορέα. Έχει πολλές, και στο φαρμακευτικό τομέα και στις μεταφορές, στα αναλώσιμα, στις νέες ενέργειες, στις νέες μορφές ενέργειας ε, για να μην ξεχάσουμε και την αεροναυπηγική με μεγάλη ε, παρουσία του Airbus και της ε, Safran σε, όλα αυτού, σε όλους αυτούς τους τομείς έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Επίσης Υπάρχει ένα μεγάλο οικονομικό πρόγραμμα με τίτλο «Ταϊλάνδη 4,0» Ε, με τομεακή προσέγγιση ιδιαίτερα ε, προγραμματισμένη. Επομένως, ε, όλες αυτές οι κινήσεις ε, βασίζονται και στην κατάρτιση. Πρέπει να πω δε ότι και η Airbus και η ε, BMW ετόλμησαν ε, να οργανώσουν κέντρα κατάρτισης στη χώρα αυτή και έχει ξεκινήσει επίσης και μια διαδικασία που αφορά την μελλοντική κατάρτιση που θα συνεχιστεί τα επόμενα χρόνια. Εμείς ήρθαμε σε επαφή με πολλούς εκπροσώπους που προβληματίζονται, εκπλήσονται από τη στάση των Ευρωπαίων γιατί τα έχουν γενικά καλές σχέσεις με όλο τον κόσμο. Είναι ε, ε, εγγεγραμμένο κατά κάποιο τρόπο στην νοοτροπία τους. Έχουν καλές σχέσεις και με την Ασία και με την Ευρώπη. Θέλουν ισορροπημένες σχέσεις με όλους. Ένας από τους ε, συνομιλητές μας μας είπε Εάν δεν κάνετε τίποτα, ε, αργότερα μπορεί στο μέλλον να γίνει ε, κινέζικο προτεκτοράτο η Ταϊλάνδη. Αυτό πραγματικά ε, μας εξέπληξε. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να υπάρχει ισορροπία στις σχέσεις με όλες τις δυνάμεις. Εν συμπεράσματι θα μπορούσα να πω ότι η Ταϊλανδία αυτή τη στιγμή θα μπορούσαν να αγνοήσουν ας πούμε την Ευρώπη και να προχωρήσουν σε διημερείς σχέσεις με μεμονωμένες χώρες ε, και ε, μέσω της αποστολής αυτής ε, κατάλαβα, κατανόησα καλύτερα αυτό που είχα πει στην ομάδα εργασίας Ευρώπης Ταϊλάνδης ότι θα πρέπει δηλαδή γρήγορα να ξεκινήσουν διερευνητικές ε, συζητήσεις ε, για μη δασμολογικές ε, διευκολύνσεις γιατί κυρίως στην αυτοκινητοβιομηχανία έχουμε νεοφυεί startup οι οποίες δουλεύουν στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας επίσης στην αεροναυπηγική αλλά και γενικότερα στην βιομηχανία γιατί εκεί η Κίνα και η Αμερική μέσω των δικών τους επιχειρήσεων ενισχύουν την παρουσία τους. Εάν χάσουμε λοιπόν υπερβολικά πολύ χρόνο δεν θα μπορέσουμε στην ε, βιομηχανία, στο βιομηχανικό τομέα γενικά να επιβάλλουμε ε, τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Τολμώ λοιπόν ε, να προτείνω στην Κομισιόν, όπως και το πρότεινα μέσω των εκεί εκπροσώπων της, να ξεκινήσουν όσο γίνεται πιο γρήγορα διερευνητικές διεργασίες έτσι ώστε να μπορέσουμε, κατά την άποψή μου, να, γίνουμε, να, να φτάσουμε σε ένα καλό επιχειρησιακό επίπεδο όταν θα φτάσουμε και θα στο εκλογές το 2019 και θα έχουν ολοκληρωθεί ε, οι εκλογικές διαδικασίες και τότε το παιχνίδι θα γίνει πολύ πιο ε, πολιτικό. Αυτά ήθελα να σας πω κύριε Πρόεδρε επαναλαμβάνοντας ότι η εντύπωση που αποκόμισα είναι ότι η Ταϊλάνδη ε, σε μια γεωγραφική περιφέρεια όπου τα πράγματα κινούνται γρηγορότερα από ό,τι σε άλλα σημεία του πλανήτη ε, είναι μια χώρα σημαντική, ενδιαφέρουσα και ως τέτοια θα πρέπει να την αντιμετωπίσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ε, David Martin was member of the... Ο David Μάρτιν ήταν μέλος της αντιπροσωπείας ε, ως μέλος της αρμόδιας επιτροπής. Ναι, ήθελα να μιλήσω, αν και συμφωνώ σε πολλά, στα περισσότερα από αυτά που ακούσαμε. Η Ταϊλάνδη δυνητικά μπορεί να αποκτήσει μεγάλη σημασία και μια ΣΕΣ με την Ταϊλάνδη θα ωφελήσει αμοιβαία τους δύο εταίρους. Δεν μπορούμε όμως να αρχίσουμε επίσημες διαπραγματεύσεις πριν από τις εκλογές και μάλιστα μέχρι και να σχηματιστεί κυβέρνηση στην Ταϊλάνδη. Αλλά συμφωνώ με τον εισηγητή ότι δεν υπάρχει λόγος να μην έχουμε τεχνικής φύσεως και άλλες συζητήσεις με τους Ταϊλανδούς ε, για να βεβαιωθούμε ότι ε, άτυπα συνεχίζονται οι τεχνικές διαπραγματεύσεις. Σε πολιτικό επίπεδο δεν μπορεί να υπάρξει συμφωνία μέχρι ότου αποκατασταθεί η ε, δημοκρατική λειτουργία. Ε, χρειάζονται βελτι... Έχουν γίνει βελτιώσεις στα εργασιακά, αλλά εργασιακά δικαιώματα, αλλά θα πρέπει να ε, υπάρξουν βελτιώσεις εις ό,τι αφορά την ελευθερία του λόγου κλπ. Ευχαριστώ. Άλλος κανείς? Κανείς. Πολύ σύντομα κύριε Πρόεδρε. Δεν είδα καμιά προετοιμασία, δεν είδα το πρόγραμμα της συνάντησης. Ε, μπορούμε να το δούμε, να διανεμηθεί. Κανένα πρόβλημα. Συνήθως το κάνουμε και θα το κάνουμε και αυτή τη φορά. Καλώς. Σχόλια από την Κομισιόν, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Να προσθέσω κάποιες παρατηρήσεις ευθυγρα... ευθυγραμμιζόμενος με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου. Γιατί τώρα είμαστε σε διαδικασία ε, επανέναρξης των συνομιλιών. Είχαμε τον Ιούλιο μια συνάντηση για θέματα εμπορίου και επενδύσεων. Είχαμε κάνει κάτι παρόμοιο την προηγούμενη χρονιά. Θα έχουμε διάλογο με το Κοινοβούλιο αργότερα, μέσα στο μήνα. Οπότε ε, γίνονται τεχνικές συζητήσεις. Επίσης μετά την ε, συνάντηση της ομάδας εργασίας τον Ιούλιο είχαμε μια πρώτη διαρευνητική συνάντηση και συζήτηση για να ξαναρχίσουμε να συζητάμε για την ΣΕΣ. Αυτό έδειξε ότι πρέπει να γίνει αρκετή δουλειά πριν μπορέσουμε να ξαναρχίσουμε αυτές τις διαπραγματεύσεις, γιατί η εμπορική πολιτική της Ένωσης έχει εξελιχθεί πάρα πολύ την προηγούμενη τετραετία αφότου ανεστάλησαν οι συνομιλίες και ίσως ό,τι αφορά το εύρος και τις διαδικασίες και τη διαφάνεια. Υπάρχουν κάποιες συζητήσεις ε, με τους Ταϊλανδούς, αλλά εκτός αυτού νομίζω ότι έχουμε τις ομάδες εργασίας ε, που συνεδριάζουν τακτικά. Δεν νομίζω περισσότερο μπορούμε να κάνουμε τεχνικές συζητήσεις ε, από ένα σημείο και μετά χωρίς να υπάρχουν και πολιτικές συζητήσεις. Οπότε θα πρέπει να ε, περιμένουμε τις εξελίξεις και τις εκλογές. Έχουν αλλάξει οι ημερομηνίε ε, των εκλογών και πριν από την Άνοιξη, για να μην σας πω το καλοκαίρι του 19, δεν θα έχει σχηματιστεί κυβέρνηση εκεί. Ε, οπότε κάνουμε κάποια προκαταρκτική διερευνητική δουλειά, αλλά έχουμε τους περιορισμούς μας και ακολουθούμε τα συμπεράσματα του Συμβουλίου. Ευχαριστώ για την πρόσθετη ενημέρωση. Κύριε Προύστ, δεν θέλει να πει τίποτε ο κύριος Προύστ. Εντάξει. Ολοκληρώσαμε λοιπόν και το σημείο 22. Και με βάση το πρόγραμμα της Επιτρόπου μπορούμε να αρχίσουμε να συζητάμε το σημείο 23 γύρω στις 11. Οπότε θα κάνουμε ένα διάλειμμα μέχρι 11 παρα 5. Uh, Αγαπητοί συνάδελφοι, χαίρομαι που έχουμε μαζί μας την Επίτροπο κυρία Μάλμστρομ που θα μας ενημερώσει για ένα καυτό θέμα. Τα αποτελέσματα της συνάντησης του Προέδρου της Κομισιόν Γιούγκερ και του Προέδρου Τραμπ σχετικά με την διαμάχη μεταξύ Ένωσης και ΕΠΑ στον τομέα του εμπορίου. Θα δώσω αμέσως το λόγο στην Επίτροπο. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη. Ελπίζω να περάσατε όμορφα το καλοκαίρι σας. Είναι ωραίο που ξαναβρισκόμαστε και που μου δίνετε τη δυνατότητα να σας ενημερώσω ε, όσο καλύτερα γίνεται μετά το καλοκαίρι για τη συνάντηση που είχαμε στο τέλος Ιουλίου. Είχα τη δυνατότητα να συνοδεύσω τον πρόεδρο Γιούγκερ στην Ουάσιγκτον στις 25 Ιουλίου. Όπως θα θυμάστε, οι ε, ε, επαφές ήταν δύσκολες όταν φτάσαμε εκεί. Εκείνη την εποχή ο πρόεδρος Τραμπ είχε χρησιμοποιήσει σκληρή ρητορική κατά της Ένωσης ε, όταν επευλήθησαν οι δασμοί για το αλουμίνιο και σε εμά και σε όλο τον κόσμο και ήταν μεγάλος ο κίνδυνος να επιβληθούν δασμοί στην αυτοκινητοβιομηχανία. Ο στόχος μας ήταν να επιδιώξουμε τον διάλογο, να αποκλιμακώσουμε την ένταση και να δούμε αν θα μπορούσαμε να ε, καταρτήσουμε ένα πιο θετικό θεματολόγιο από αυτό που ε, κλιμακωνόταν. Γιατί εμείς ε, στο χάλιβα και το αλουμίνιο αντιδράσαμε με αντίπεινα και ετοιμάζαμε και κατάλογο πιθανών αντίμετρων εάν οι δασμοί ε, επιβάλλονταν για τα αυτοκίνητα και τις εξατμίσεις. Αυτό προετοιμαζόταν, υφίστατο λοιπόν το θέμα και αν χρειαζόταν θα το εφαρμόζαμε. Μία διαμάχη για τους ε, δασμούς στα αυτοκίνητα θα είχε τεράστιες επιπτώσεις στην αυτοκινητοβιομηχανία, όχι μόνο στις χώρες που παράγουν αυτοκίνητα, αλλά και σε άλλες χώρες. Και η επιβολή δασμών θα επηρέαζε ε, τις εξαγωγές κατά 51 δις. Πολύ, πολύ μεγάλο ποσό δηλαδή. Είχαμε επικοδομητική συζήτηση με τον πρόεδρο Τραμπ και την ομάδα του, γιατί παρευρέθησαν και αρκετοί υπουργοί στο Λευκό Οίκο και φτάσαμε σε μια πολιτική συμφωνία να δημιουργήσουμε εκτελεστική ομάδα εργασίας η οποία θα προσπαθούσε να εργαστεί επί θετικού θεματολογίου. Αυτή η εκτελεστική ομάδα εργασίας ε, θα ήταν ε, με επικεφαλή σε μένα και τον ε, Υπουργό Λάιτ Λάιτνερ και το καλοκαίρι οι ομάδες μας ε, συναντήθηκαν για να προετοιμάσουν τα σχετικά. Αποφασίσαμε ότι θα διερευνούσαμε τις δυνατότητες ε, εμπορικής συμφωνίας που θα εστιάζει σε βιομηχανικά αγαθά. Είπαμε ότι είμαστε έτοιμοι να ε, πάμε σε μηδενικούς δασμούς όλα τα βιομηχανικά αγαθά αν κάνουν το ίδιο και οι ΙΠΑ, δηλαδή αυτό θα λειτουργούσε σε βάση αμοιβαιότητας και ότι θα περιοριζόμαστε σε βιομηχανικά αγαθά. Η Γεωργία δεν θα ε, ήταν στη συμφωνία ούτε οι δημόσιες συμβάσεις ως έχουν σήμερα. Θα ήταν μικρότερη αλλά σημαντική συμφωνία με την έννοια ότι θα ήταν αμοιβαία υποφελής και για την Ένωση και για τις ΕΠΑ. Συμφωνήσαμε επίσης σε αυτά τα πλαίσια να διευκολύνουμε την ενεργειακή συνεργασία. Σήμερα περιπλέκεται για χώρες που θέλουν να εισάγουν αέριο από τις ΗΠΑ, είναι δύσκολο να πάρουν τις άδειες, αυτό είναι κάτι που κάθε κράτος μέλος το αποφασίζει μόνο του, αλλά αν θέλουν να κάνουν εισαγωγές αερίου από τη ΣΥΠΑ είναι περίπλοκο το θέμα. Στα πλαίσια μιας τέτοιας συμφωνίας θα διευκολύνεται η αδειοδότηση στις χώρες που θέλουν να κάνουν εξαγωγές. Ε, αυτό ήταν ένα κομμάτι της διαπραγμάτευσης. Το άλλο κομμάτι είναι, ήταν να δούμε αν μπορούσαμε να συνεργαστούμε σε εθελοντική βάση εκτός συμφωνίας επί ορισμένων θεμάτων σχετικά με τα πρότυπα στα χημικά, ιατρικά προϊόντα, φαρμακευτικά προϊόντα. Ήδη είχε γίνει πολύ προπαρασκευαστική δουλειά και θέλαμε να διερευνήσουμε να δούμε τι μπορεί να γίνει. Κάποια θέματα ήταν εύκολα, δεν ήταν περίπλοκα, αλλά είναι πιο περίπλοκα και εκεί εστιάζουμε και να δούμε πού μπορούμε να επιτύχουμε γρήγορα αποτελέσματα. Επίσης συμφωνήσαμε και το είδατε αυτό στην δήλωση ε, των δύο προέδρων ότι στο βαθμό που συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις συμφωνούν οι δύο πλευρές ότι δεν θα επιβληθούν νέοι δασμοί και οι υφιστάμενοι δασμοί θα επαναξιολογηθούν. Ο στόχος είναι προφανώς στα πλαίσια των εργασιών που θα πάρουν πιο συγκεκριμένη μορφή, ο στόχος είναι να, να, πείσουμε τις είπα να καταργήσουν τους δασμούς στο αλουμίνιο και το χάλιβα. Και αν συμβεί αυτό, θα είμαστε έτοιμοι και εμείς να καταργήσουμε ε, τους δασμούς από την πλευρά μας. Ε, Συμφωνήσαμε επίσης να συνεργαστούμε στενά μεταξύ μας και να ενημερώσουμε και τον ΠΟΕ σχετικά με τις αθέμητες εμπορικές πρακτικές ε, όπως ε, ε, πλεονάζουσα ε, παραγωγική δυνατότητα, αναγκαστική, εξαναγκαστική μεταφορά τεχνολογιών, ε, κακόβουλες πρακτικές, ε, κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας, υπερπροσφοράς. Κάναμε συναντήσεις για προτάσεις επί νέων κανόνων στα πλαίσια του ΠΟΕ. Προφανώς χρειάζονται και οι άλλοι να συμμετάσχουν. Αν όμω η ίπα, η Ένωση και η Ιαπωνία παρουσιάσουν προτάσεις, αυτό θα είναι πολύ σημαντικό. Και αυτό είναι σημαντικό αποτέλεσμα σε σχέση με την μεγάλη πρόκληση μπροστά μας, δηλαδή να ενισχύσουμε το σύστημα που στηρίζεται σε κανόνες. Αυτή η διαδικασία άρχισε και αργότερα σε πλαίσιο τριμερές υπήρξε επιβεβαίωση από τον πρόεδρο Τραμπ και τον πρόεδρο Γιούγκερ. Επιβεβαιώθηκε ε, ε, η συνέχιση. Ε, προχωράμε με πνεύμα εμπιστοσύνη. Θέλουμε να δημιουργηθούν οι απαραίτητε δομέ. Δεν υπάρχουν χρονοδιαγράμματα, αλλά προφανώ θέλουμε η πρόοδο να είναι όσο γίνεται πιο γρήγορη. Είπαμε σαφώ ότι δεν διαπραγματευόμαστε με το πιστόλι στον κρόταφο. Αυτό είναι σημαντικό επί της ουσίας, εκεί εστιάζομαι. Ε, η εκτελεστική ομάδα εργασίας έχει πολιτική εντολή και θα παρουσιάσουμε συστάσεις σχετικά με το πώς θα προχωρήσουμε. Αφού γίνει αυτό, πριν αρχίσουμε τις πραγμα... πραγματικές ουσιαστικές διαπραγματεύσεις, θέλουμε εντολή από τα κράτη-μέλη. Πρόκειται για μια πρώτη διαρευνητική διαδικασία που άρχισε ήδη, όπως είπα, το καλοκαίρι και θα συνεχιστεί τις πρώτες εβδομάδες του Σεπτεμβρίου. Αυτή είναι μια ευκαιρία που έχουμε να συνεργαστούμε με τους Αμερικανούς εταίρους για να αντιστρέψουμε ε, την κατάσταση, το οφείλουμε στους πολίτες, να βρούμε μια θετική ατζέντα για να συνεχίσουμε και να ξεπεράσουμε τα προβλήματα που είχαμε στην αρχή του καλοκαιριού όπου κλιμακωνόταν η ένταση καθημερινά. Αυτά. Προς το παρόν, κύριε Πρόεδρε, προφανώς θα συνεχίσω να ενημερώνω τα μέλη της Επιτροπής σας. Τώρα είμαι έτοιμη να απαντήσω τυχόν ερωτήσει σας Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Επίτροπε. Αλλάζω τίτλο και ως απλός ε, εισηγητής για τις σχέσεις ΕΠΑ Ευρωπαϊκής Ένωσης θα θέσω μερικά ερωτήματα στα γερμανικά. Κυρία Επίτροπε, Αναφέρομαι στην τελευταία σας παρατήρηση που τη βρίσκω σημαντική. Δηλαδή ότι τώρα γίνονται συνομιλίες ξανά, είναι μεγάλη επιτυχία αυτή σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο όπου έχουμε παγκόσμιες αλυσίδες αξίας, ένας εμπορικός πόλεμος δεν έχει κανένα νόημα. Ε, ε, αντίθετα, καταστρέφει τις αλυσίδες αυτές και υπονομεύει τα συμφέροντα όλων. Είναι λοιπόν θετικό δείγμα η σύνοδος, η συνάντηση κορυφής που αναφέρατε. Έχω να κάνω πέντε παρατηρήσεις κάπως, που, που αξιολογούν κάπως κριτικά το αποτέλεσμα. Πρώτον, πάντα λέγαμε ότι δεν θέλουμε να κάνουμε παραχωρήσεις στο βαθμό που οι κρατικοί δασμοί για το χάλιβα υφίστανται και υπάρχει και η απειλή ε, επιβολής δασμών κατά, ε, ε, στα αυτοκίνητα. Αυτό εξακολουθεί να υπάρχει, δηλαδή είναι ενισχύει η δασμή στο χάλιβα και το αλουμίνιο και η απειλή για τα αυτοκίνητα δεν έχει εξαλειφθεί διότι έχουν ε, συμπεριληφθεί σε μια πιθανή διαπραγματευτική εντολή για τα, διαπρα... βιομηχανικά αγαθά. Και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό για το Κοινοβούλιο. Δηλαδή, μην κάνουμε παραχωρήσεις προτού δώσουν οι ΙΠΑ σαφή δείγματα ότι ε, θα παρατηθούν από, αυτή τη δυνατότητα που έχουν επιβολή των δασμών. Δεύτερον, οι ΙΠΑ ε, επικεντρώθηκαν μόνο στους δασμούς. Κυρία Επίτροπε, τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων του ΠΟΕ για τους δασμούς ε, ήδη αποτελούν κομμάτι διεθνούς συμφωνίας. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν γιατί ο πρόεδρος ε, τον είπα το θεωρεί αυτό άδικο. Αφού συμμετέχουν στον ΠΟΕ και άλλα θέματα που είναι σημαντικά για μας όπως το ζήτημα των υπηρεσιών, των δημοσίων προμηθειών, συμβάσεων όλα αυτά δεν λαμβάνονται υπόψη. Θυμίζω πάλι ότι η ΕΠΑ έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν πλεόνασμα 50 δις πέρσι στον τομέα των υπηρεσιών και 80 δις ε, πήραν για ε, άδειες ε, και διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Αυτό ήταν το ενδιαφέρον στην ίδρυση του ΠΟΕ. Όχι τόσο οι δασμοί, αλλά οι άλλοι τομείς. Και αυτό δεν ε, συζητήθηκε. Τώρα, η συνεργασία για τα πρότυπα είναι πολύ σημαντική. Ε, εγώ ασχολήθηκα στα πλαίσια του TTIP ακριβώς με αυτό το θέμα. Αλλά υπάρχουν προβλήματα εδώ γιατί υπάρχουν διαφορετικά πρότυπα και λόγω ανταγωνισμού αλλά και λόγω των διατάξεών μας ε, για την προστασία των καταναλωτών και τις υπηρεσίες γενικού ε, συμφέροντος. Γιατί λοιπόν εμείς θα πρέπει να παρεκκλίνουμε από τις ευρωπαϊκές ε, θέσεις, εκτός και αν υπάρχουν απτές πρόοδοι. Χρειάζεται μεταρρύθμιση του ΠΟΕ. Προφανώς θέλουμε να προχωρήσουμε και τα τρία αυτά. Το θέμα των αρμοδιοτήτων του ΠΟΕ, της, ε, των δικαιοδοτικών οργάνων του, ε, την λειτουργικότητα και αποτελεσματικότητα το που έπρεπε να τα δούμε. Αλλά δεν θέλουμε να στραφούμε ενάντια σε έναν άλλον εταίρο του ΠΟΕ. Θα πρέπει τα συμφέροντά μας να τα ε, διασφαλίσουμε στα πλαίσια της μεταρρυθμιστικής διαδικασίας του ΠΟΕ. Και η ΥΠΑ τη Δευτέρα δήλωσαν ότι έναν δεν θα δεχτούν επαναδιορισμό δικαστή στο δικαιοδοτικό όργανο αυτό, θέτει σε ε, ε, αμφιβολία ε, την αποτελεσματικότητα και δεν προωθεί την εμπιστοσύνη. Επίσης, η στρατηγική του κυρίου Τραμπ, διέρη βασίλευε, δεν μπορεί να οδηγήσει σε επιτυχία. Δηλαδή, ο Σόζον ε, αυτόν σωθήτο είναι η πολιτική ψάχνουν για ειδικέ αγορέ. Εμείς θέλουμε μια σαφή κοινή ευρωπαϊκή θέση για προσέγγιση βασισμένη σε κανόνες και αυτή την πολιτική και αυτές τις αξίες θα πρέπει να τις καταστήσουμε σαφέστατες. Αυτά από την πλευρά του Μπέρντ Λάγκε ως εισηγητή. Και τώρα ε, τα μέλη σκιώδεσε. Η κυρία Κουιστούτ Βορόβολε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Επίτροπε για την ε, επίσκεψή σας εδώ. Ζητώ συγγνώμη που καθυστέρησα, αλλά έκανα συνομιλίες ε, με το Μαρόκο για την Δυτική Σαχάρα, που είναι και αυτή ένα περίπλοκο θέμα. Και με συγχωρείτε. Θα ήθελα λοιπόν να περάσω στην πρώτη μου ερώτηση. έχουμε ένα καθημερινά μεταβαλλόμενο κόσμο και ε, ε, προβλήματα παντού. Εμείς ως, αναρωτιέμαι, ως Ευρωπαϊκή Ένωση ακολουθούμε μια συγκεκριμένη στρατηγική που μας ε, ε, καθιστά ορατούς όλα αυτά τα θέματα. Μιλάμε για τις αξίες μας, τα πρότυπά μας που θέλουμε να τα διατηρήσουμε, θαυμάσια όλα αυτά αλλά τα θεωρώ και λίγο μη ρεαλιστικά. Και το λέω ειλικρινά, μιλάω ανοιχτά. Ο κόσμος, όπως σας είπα, αλλάζει συνεχώς. Πρέπει να προσέξουμε να μην απομονωθούμε στο τέλος. Αυτό το λέω και εκ από την, την πείρα που έχω αποκομίσει από την Κεντρική Ασία. Είναι λοιπόν ένα κεντρικό ερώτημα. Δεν πρέπει κάποια πράγματα στην εμπορική μας πολιτική να τα τοποθετήσουμε σε διαφορετική βάση. Δεύτερη ερώτηση. Προφανής ερώτηση νομίζω. Πώς μπορούμε να προχωρήσουμε στις σχέσεις μας με τις ΗΠΑ όταν καθημερινά έρχεται διαφορετική μια διαφορετική δήλωση. Εντάξει, να είμαστε ευέλικτοι, αλλά ανάλογα με τον Αμερικανό συνομιλητή είναι και διαφορετικό το μήνυμα που φτάνει και ε, δεύτερον μπορεί την επόμενη μέρα να αλλάξουν όλα. Έχει συμβεί αυτό. Πώς μπορούμε έτσι να διαπραγματευτούμε, είναι ένα ένιγμα αυτό για μένα. Τρίτον, στην αυτά, αν ισχύουν αυτά που ακούσαμε, ο Καναδάς είναι ε, λίγο απομονωμένος από τους εταίρους του. Αυτό θα έχει επίδραση στη Συμφωνία ΣΕΤΑ. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Επίτροπο και εγώ. Ε, καλή επάνωδο και ε, εύχομαι να εργαστείτε καλά τους επόμενους μήνες. Πρώτα απ' όλα θα κάνω κάποιες σκέψεις σχετικά με το γεγονός ότι ε, τουλάχιστον ε, σταμάτησε η κλιμάκωση μέσω αυτής της ε, συνάντησης και εγώ προσωπικά θα ήθελα να υπογραμμίσω κάποιες από τις παρατηρήσεις που έκαναν οι προαλήσαντες συνάδελφοι. Πρώτα απ' όλα το Executive Working Group που ήταν ένα από τα αποτελέσματα της ε, ε, διάλεξης. Ε, υπενθυμίζω σε όλους ότι το Κοινοβούλιο θέλει και πρέπει να συμμετάσχει στη διαδικασία. Το υπενθυμίσατε κι εσείς. Για μένα είναι σημαντικό να γνωρίζουμε όλα τα στοιχεία έτσι ώστε να μπορούμε να παρακολουθούμε βήμα προς βήμα όλα τα στοιχεία της εντολής που έδωσαν τα κράτη-μέλη και το Κοινοβούλιο να είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με όλη τη διαδικασία γιατί υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία απορρέουν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και που είναι σημαντικά. Δύο δύο στοιχεία. Πρώτον, όσον αφορά ε, τον τρόπο μηχανισμό λειτουργία του Διεθνούς Φόρουμ, παραμένει αυτή η τεράστια αμφισημία της στάση των Ηνωμένων Πολιτειών που προσπαθεί να ε, μπλοκάρει ε, την διαδικασία με το να μην διορίζει την δικαστή και αυτό βεβαίως είναι στοιχείο το οποίο οπωσδήποτε πρέπει να ληφθεί υπόψη στις συζητήσεις με τον εταίρο δεύτερο στοιχείο που θέλω να αναφέρω είναι η στάση των Ηνωμένων Πολιτειών όσον αφορά την συμμετοχή στη Συμφωνία των Παρισίων και οτιδήποτε σχετίζεται με τις εργασίες που συνεχίζουν ε, την περιβαλλοντική εργασία και την εργασία για την κλιματική αλλαγή. Αυτό αποτελεί τεράστιο εμπόδιο ε, όσον αφορά την δυνατότητα καρποφόρου διαλόγου ε, με την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να ασκήσουμε πίεση για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε την εργασία. Τελευταίο στοιχείο ή μάλλον ερώτηση. Σήμερα το πρωί αλλά και τις προηγούμενες μέρες Ακούσαμε διάφορα στοιχεία ότι δηλαδή καταγράφεται ε, αρχή τροποποίησης της τάσης ε, της ε, κυβέρνησης Τραμπ λόγω των πιέσεων των Αμερικανών εργαζομένων που πλέον λένε αυτό που εμείς πάντα λέγαμε εξ αρχής δηλαδή ότι το θέμα των δασμών εν τέλει θα στραφεί εναντίον των Αμερικανών εργαζομένων. Να δούμε πώς είναι δυνατόν να βοηθήσουμε και λαμβάνοντας λαμβάνοντας υπόψη αυτό το στοιχείο την διαδικασία η οποία στόχο θα έχει την γενική βελτίωση μιας εργασίας που προς ώρας μας φαίνεται ακόμα πολύ περίπλοκη γιατί όπως έλεγε και εσάς προηγουμένως η αμφισημία με την οποία εργάζεται και ε, ε, ομιλεί και ο πρόεδρος Τραμπ είναι διαρκής. Ευχαριστώ. Ο ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κυρία Επίτροπε που ήρθατε. Το θέμα είναι καυτό στην κοινή γνώμη. Πρέπει να κάνουμε κάποιες κριτικές ερωτήσεις. Καταρχήν δεν έχετε εντολή για τις διαπραγματεύσεις. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το Μάιο και τον Ιούλιο είπατε και ο πρόεδρος Γιούγκερ το είπε ότι μετά το πάγωμα του TTIP ε, πρέπει να υπάρχει εντολή του Συμβουλίου. Δεν βλέπω και ενιαία θέση των κρατών μελών. Βλέπω τον Γάλλο Υπουργό Οικονομικών, τον Γερμανό ομολογό του. Βλέπουμε να διήστανται οι απόψεις. Δεν είπατε όχι διαπραγματεύσεις με το πιστόλι στο Γκρόταφο. Ε, πρέπει λοιπόν να συνεννοηθούμε. Η συνάδελφος Μόσκα έχει δίκιο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιμένει με βάση την εμπειρία του παρελθόντος να μπορούμε να έχουμε λόγο και εμείς στις διαδικασίες. Οι μελλοντικέ, διατλαντικές σχέσεις και συνεργασία στο εμπόριο ε, και στην οικονομία πώς θα είναι. Αν η πρόθεση είναι να περιοριστεί συμφωνία στα βιομηχανικά αγαθά, τι θα γίνει με τα κοινωνικά πρότυπα, τα περιβαλλοντικά πρότυπα. Ε, στη διαδικασία TTIP φάνηκε ότι οι πολίτες ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, θα υποστούν ζημία. Τι θα γίνει με τη σόγια, τι θα γίνει με την ενδεχόμενη εισαγωγή της. Ε, επίσης, τι θα γίνει με τις εμπορικές σχέσεις είπα Κίνας ε, και πώς θα επηρεαστούν οι εξαγωγές. Θέλουμε να δούμε το ευρύτερο πλαίσιο και καλό είναι να έχουμε συγκεκριμένα αιτήματα που θα έχουμε διατυπώσει προς τον πρόεδρο Τραμπ ε, για να μην ε, ε, είμαστε εκτεθειμένοι και να κινδυνεύουμε από τις μεγάλες πολυεθνικές. Και χρειάζεται συνεργασία και με τα μέλη του ΠΟΕ για τη μεταρρύθμιση του τελευταίου. Μαρία Ρένα. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι με μεγάλη έκπληξη διαπιστώσαμε στη άκρη των διακοπών τα όσα ε, συμβαίνουν. Κυρία Μάλστρομ, μα λέτε ότι ε, δεν δέχεστε, ε, μα είχατε πει δεν δέχεστε να διαπιστώνετε, να διαπραγματεύεστε, συγγνώμη, υπό την απειλή, αλλά φαίνεται ότι δεν είναι η ίδια γνώμη του Προέδρου Γιούνκερ. Θα ήθελα λοιπόν να σα ρωτήσω ποιο είναι το καθεστώ αυτή τη διαπραγματεύση κάθε φορά που σα ρωτούμε, έτσι ώστε να βάλετε νέες διατάξει σε στην δια, ε, διαπραγμάτευση, λέτε «Α, δεν έχω τέτοια εντολή». Ε, εδώ πάλι μας λέτε ε, δεν έχετε όμως καμία δυσκολία να διαπραγματευτείτε κάτι το οποίο όμως είναι εκτός ε, της εντολής. Δεύτερη ερώτηση. Ο κύριος Ελμάγερ ως τι και υπό ποια λειτουργία είχε την θέση του επικεφαλής διαπραγματευτή. Ποιο ήταν ο πραγματικός ρόλος, ο επίσημος ρόλος αυτού του κυρίου στις διαπραγματεύσεις. Τρίτη ερώτηση, το είπατε κι εσείς, δεν διαπραγματευόμαστε υπό απειλές. Τι γίνεται λοιπόν όσον αφορά το θέμα των δασμών και όσον αφορά ε, το, ε, ε, την επεμπλοκή των Ηνωμένων Πολιτειών όσον αφορά την πολυμέρεια. Έχουμε την εντύπωση ότι εδώ έχουμε μια διαπραγμάτευση όπου κρατάει κρυμμένα χαρτιά και έχει όλα τα του με την πλευρά του ο πρόεδρος Τραμπ σε αυτήν την διαπραγμάτευση. Ναι, είδαμε την επικριτική στάση των πολιτών όσον αφορά την συμφωνία TTIP. Είδαμε ότι ε, ε, δεν υπήρχε καθόλου διαφάνεια στη διαδικασία. Εδώ βλέπουμε μια διαδικασία διαπραγμάτευσης ε, η οποία δεν έχει επίσης καμία διαφάνεια και αυτό πρέπει οπωσδήποτε να εξηγηθεί στους πολίτες που επικριτικά τη βλέπουν. Ευχαριστώ πολύ. Πολλοί το είπαν, αλλά και εγώ θέλω να εκφράσω την απορία μου πώς μπορούν να αρχίζουν έτσι οι συνομιλίες. Γιατί ακόμα δεν διαπραγματευτήκαμε και ήδη κάναμε πολλές παραχωρήσεις προς τις είπα, ενώ εκείνοι δεν είπαν καν ότι θα αποσύρουν τις απειλές. Είπαν θα το δούμε, θα το δούμε. Δηλαδή εξακολουθούν οι απειλές και επίσης ο γεωργικός τομέας που δεν έχει ε, γίνει αντικείμενο των διαπραγματεύσεων. Ποια είναι η μακροπρόθεσμη στρατηγική μας. Δηλαδή με αυτή τη στάση τι θα επιτύχουμε. Θα επιτύχουμε να γίνουμε υποχείρια του Τραμπ, ο οποίος προσπαθεί να διχάσει τον κόσμο, να ασκήσει πιέσεις και να κάνει υποφελείς συμφωνίες για τις ΣΥΠΑ. Και εμείς εξυπηρετούμε αυτή την πολιτική του με αυτόν τον τρόπο. Γιατί ε, δεν είναι αντικείμενο συζήτηση στα σημαντικά. Μιλάμε για θέματα που ωφελούν τη ΣΥΠΑ. Αυτό είναι το αντίθετο από αυτό που έλεγε μέχρι τώρα η Κομισιόν και αυτό που με ενδιαφέρει πάνω απ' όλα. Τι πρέπει να λέει η διαπραγματευτική εντολή. Όχι να λέει μόνο αυτά που θέλουν οι ΙΠΑ. Έχετε σκεφτεί τι θα πούμε εμείς, πώς, τι μορφή θα έχει η διαπραγματευτική εντολή. Γιατί είπατε ότι κάποια στιγμή θα συσταθεί μια εντολή. Κανονικά γίνεται πριν από τι συνομιλίε κάτι τέτοιο, αλλά τέλος πάντων. Με ενδιαφέρει όμως το περιεχόμενο της διαπραγματευτική εντολής. ECR, Εμαλάκη. Κύριε Επίτροπε, οι συναδελφοί κάλυψαν τα περισσότερα, εξεπλάγημεν όμως όλοι το καλοκαίρι με αυτά που έγιναν. Ο στόχος ε, του Τραμ και των ΗΠΑ είναι μηδέν παντού σε δασμούς και μη δεσμολογικά εμπόδια. Υπάρχει εμπόδιο με Υπάρχει χρονοδιάγραμμα γι' αυτά. Πότε μπορεί να επιτευχθεί αυτό. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Αν Μαρή Πρόεδρε. 20 Μαΐου στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μιλήσαμε για τους δασμούς για χάλιβα και αλουμίνιο. Κύριε Μάλστρομ είχε πει τότε ότι χρειαζόμαστε εντολή το οποία θα δώσει το Συμβούλιο στην Κομισιόν για να διαπραγματευτεί. Ερώτημα πρώτο. Ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις. Είχε εντολή η Κομισιόν από το Συμβούλιο. Και αν ναι, ποια εντολή. Επίσης, Όλοι είπαμε ότι η Συμβουλή Κομισιόν και ο κόσμος θεωρήσαν ότι η TTIP είναι απαράδεκτη. Και τώρα βρισκόμαστε όμως ξανά με τον πιστόλι στον κρόταφο. Και ξέρουμε ότι οι συνομιλίες για την ε, TTIP δεν είναι σε καθεστώ διαφάνεια. Τι γίνεται με τους στόχους για τη μεταβολή του κλίματος και που πάμε ως προς το στόχο μηδέν σε δεσμούς και μη δεσμολογικά εμπόδια. Και αν αυτό το πετύχουμε, με βάση ποια εντολή ο πρόεδρος Γιούνκερ έκανε, τις δηλώσεις που έκανε. Θα δεχθούμε εισαγωγές σόγες όταν Ξέρουμε ότι το 90% της σόγιας είναι γενετικώς τροποποιημένη. Επίσης, ο τομέας των μεταφορών που επιβαρύνει τα μάλλα το περιβάλλον. Και επίση τη μέτρα σκοπεύει να λάβει η Κομισιόν για να σταματήσει τις εισαγωγές γενετικώς τροποποιημένης σόγιας. Και γιατί να εισάγουμε υγροποιημένο φυσικό αέριο, να ξέρουμε ότι στην ε, Ηνωμένε Πολιτείε παράγεται πώ το λιθό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Δύο από τα ερωτήματά μου ήδη ετέθησαν, δεν θα τα επαναλάβω προφανώ. Αλλά θυμίζω, δεσμού στην αυτοκινητοβιομηχανία και υποθέσει των ΠΟΕ. Ήσασταν ε, πάρα πολύ σύντομο. και ευχαριστώ, είμαι χωρίς μικρόφωνο, η μιλήτρια. Ευχαριστώ πολύ κυρία Επίτροπε ε, για την παρουσία σας σήμερα εδώ. Πιστεύω ότι πραγματικά η κατάσταση είναι καλύτερη από αυτήν που αντιμετωπίζαμε τον Ιούνιο, διότι ε, η ε, διαδικασία ενός εμπορικού πολέμου δεν ευχαριστεί κανέναν και οπωσδήποτε και αμφισβήτητα πάντα ο διάλογος είναι καλύτερος. Ωστόσο παραμένουν δύο ζητήματα τα οποία αφορούν τους όρους και συνθήκες ε, της διαπραγμάτευσης και τη συνέχεια της διαπραγμάτευσης. Ε, Υπάρχει από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης εμπορική πολιτική η οποία δεν προσπαθεί μόνο να βελτιώσει τις ε, συνθήκες ε, ε, και τις αξίες των εμπορικών συμφωνιών αλλά και να εξάγει αυτές τις αξίες και συνθήκες. Δυστυχώς ο πρόεδρος Τραμπ έχει ένα δικό του τρόπο δράσης και αυτού του τρόπου υπεραμείνεται φυσικά. Και δεν είναι ο ίδιος τρόπος με τον οποίο κάνουμε τα πράγματα εμείς εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν κάνει κανείς έναν ε, διάλογο τόσο περίπλοκο, αφήνοντας απ' έξω εμπορικά θέματα, όπως ας πούμε δημόσιες ε, ε, συμβάσεις, που είναι τόσο σημαντικές, και θέματα τα οποία αφήνονται απ' έξω όπως ας πούμε αυτό που σας λέω η πρόσβαση στις αγορές αυτές για των δημοσίων προμηθειών ήδη μας προβληματίζει και εγώ αναρωτιέμαι εμείς και το είπατε κι εσείς, λέμε ότι δεν είναι δυνατόν ε, να έχουμε ε, διαπραγματεύσεις ε, υπό τις απειλές για τα αυτοκίνητα αλλά και δασμολογικό πόλεμο για το χάλιβα, αλλά από την άλλη μεριά κάνουμε πολλές υποχωρήσεις. Εγώ νομίζω ότι το να δεχτούμε κάποιες αρχές οι οποίες ας πούμε ε, είναι επιζήμιες ε, για τις ε, βρόσιμες ελιές και από την άλλη πλευρά να μην κάνουμε κάποια, να μην, να μην ζητούμε από τις, Ευρωπα... από τις Ηνωμένες Πολιτείες μια κίνηση η οποία να δείχνει ότι και αυτό τι ε, κάνει κάποια υποχώρηση δεν είναι σωστή. Επίσης ε, θα υπάρξει κεφάλαιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη, γιατί εμείς πάντα λέγαμε ότι πρέπει να υπάρχουν τέτοια κεφάλαια για τη βιώσιμη ανάπτυξη και δεν καταλαβαίνω γιατί αυτό δεν αναφέρεται καθόλου, γιατί εδώ δεν ε, μιλάμε μόνο για τον τρόπο με τον οποίο θα ανταλλάσσουμε προϊόντα, αλλά και με ποιο τρόπο θα ανταλλάσσουμε τα προϊόντα. Έχουμε εδώ απέναντί μας ένα ομιλητή ο οποίος έχει αποφύγει από τη Συμφωνία ε, των Παρισίων. Ε, δεν ε, προσπίζεται την ειρήνη, δεν προσπίζεται την ισότητα των φίλων. Ξέρουμε με ποιο τρόπο αντιμετωπίζει και φέρεται στις γυναίκες. Πώς είναι δυνατόν όλα αυτά τα θέματα να τα παραβλέψουμε στη Συμφωνία. Ευχαριστώ. Γουίδο Σίλβα Περέιρα. Obrigado, Presidente. Senhora Comissária, primeiro um ponto político. Κυρία Επίτροπε, ε, θα ήθελα να κάνω μια πολιτική φύσεως παρατήρηση πρώτα απ' όλα. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή ε, ε, ε, δέχονται επίθεση από την ε, κυβέρνηση Τραμπ και από τον ίδιο τον πρόεδρο. Πρώτα σταμάτησε τις διαπραγματεύσεις, μετά τον πόλεμο για το αλουμίνιο και μετά απειλές για την αυτοκινητοβιομηχανία. Επίσης πολιτικά μηνύματα τα οποία αποδυναμώνουν την Ατλαντική συνεργασία όσον αφορά τους τομείς ας πούμε της ε, ε, άμυνας, επίσης αυτή η υποστήριξη στο Brexit κλπ. Απέναντι σε μια τέτοια κατάσταση, κυρία Επίτροπε, δεν είναι δυνατόν εμείς να δώσουμε ακόμα μια νίκη ή έστω και μια αυταπάτη νίκης στην ε, διοίκηση Τραμπ. Το Κοινοβούλιο ε, οποτεδήποτε ε, αναφέρεται σε ε, προγράμματα ή σε προτάσεις εμπορικού πολέμου πάντα είχε μια συγκεκριμένη αντιμετώπιση. Εγώ νομίζω ότι πραγματικά ε, θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τα λάβει υπόψη τη όλα αυτά, να λάβει υπόψη τη και όσα λέει κατά διαστήματα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ρωτώ λοιπόν, ποιο είναι ο πραγματικό στόχο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μπορούμε να πούμε τώρα ότι έχουν ξαναρχίσει οι διαπραγματεύσει τη TTIP, γιατί οι διαπραγματεύσει με τι ε, Ηνωμένε Πολιτείε για του ε, για, μηδενικού δασμού και για μηδενικού εμπορικού φραγμού δεν μπορούν μπορούν παρά να ειδωθούν σε ένα ευρύτερο πλαίσιο των, ε, αυτό των ε, ευρύτερων ε, σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών. Πώς προτίθεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έχει την δημοκρατική νομιμοποίηση για αυτήν την σχέση η οποία πλέον αντιμετωπίζει προβλήματα. Ευχαριστώ. Um, Ευχαριστώ. Τρεις απλές ερωτήσεις. Πρώτον, κάποιοι τομεί όπω η αυτοκινητοβιομηχανία βαρύνονται με δασμού περισσότερου ει βάρο των ΗΠΑ παρά ει βάρο τη Ευρώπη. Η Κομισιόν έχει σχέδια να μειώσει αυτού του δασμού στα αμερικανικά αυτοκίνητα, ώστε οι δασμοί εκατέρωθαν να είναι οι ίδιοι. Και αν όχι, εκτιμώ ότι τα σχόλια, πολλά από τα σχόλια των συναδέλφων είναι ανεδαφικά. Δεύτερον, εμείς εξάγουμε περισσότερα στη ΣΥΠΑ από ότι αντιστρόφως. Περισσότερα κατά 150 περίπου δισεκατομμύρια. Είναι περίπου το ΑΕΠ της Ουγγαρίας, συνειδητοποιείτε. Κατά τη γνώμη σας και κατά τη γνώμη της Κομισιόν εν γέννη, ε, αυτό είναι μια βιώσιμη κατάσταση μπορεί να συνεχιστεί. Και τέλος, μια γενικότερη ερώτηση. Η Γερμανία με αξιοθαύμαστο τρόπο θα έλεγα εξασφάλισε ένα εξαιρετικό εμπορικό πλέον με 7,6% του ΕΠ, παρακαλώ. Κατά τη γνώμη της Κομισιόν αυτό είναι μια βιώσιμη κατάσταση και είναι κάτι το οποίο επιτρέπεται να συνεχιστεί. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, πολύ ωραία. Δεν έχω άλλα για τον λόγο που η Επίτροπος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι βουλευτές. Ίσως δεν ήμουν σαφή στην αρχή, κάποιοι καθυστέρησαν κιόλας, αλλά με δεν διαπραγματευόμαστε τίποτα. Έχουμε μια ομάδα εργασία απλώς. Τίποτα άλλο. Έχουμε σοβαρότερες διαφωνίε με τις ΗΠΑ στην εμπορική πολιτική και σε άλλες πολιτικές. Δεν συμφωνούμε με τι ενεργειές τους στον ΠΟΕ. Δεν συμφωνούμε με την ε, αντίσταση που παρουσιάζουν στον διορισμό δικαστή. Σε μερικού τομεί προσπαθούμε να βρούμε λύσει μαζί τους, μαζί με τις ΗΠΑ και μαζί με άλλες χώρες στον ΠΟΕ για να δούμε αν υπάρχει όντω διέξοδος και συνεργαζόμαστε και με άλλε χώρες, καμιά φορά και τριμερό με τη ΣΥΠΑ, με την Ιαπωνία στον ΠΟΕ, για να δούμε πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τους υφιστάμενους κανόνες. Και εδώ όλοι συμφωνούμε νομίζω, γιατί ότι όλοι συμφωνούμε ότι χρειαζόμαστε νέους κανόνες στον ΠΟΕ, χρειαζόμαστε ένα νέο ΠΟΕ. Μιλήσαμε με τι ΗΠΑ, την Ιαπωνία, μιλάμε και με την Κίνα. Προφανώς πρέπει να συμμετάσχει η Κίνα, γιατί πολλά από τα προβλήματα απορρέουν από τη στάση της Κίνας και πρέπει να σας πω ότι πολλοί συμφωνούν με εμάς τον ΠΟΕ, με, μαζί με τους οποίους κατεβάζουμε προτάσεις και ελπίζω ότι κάποια στιγμή θα παρέλθουμε και θα το ξανασυζητήσουμε με περισσότερες λεπτομέρειες. Διαφωνούμε με την επιβολή δασμών με τη ΣΥΠΑ ο Χάλιβας και το λουμίνιο βαρύνονται με δασμούς που για μας είναι παράνομοι. Δεν συνάδουν με τους κανόνες του ΠΟΕ, ούτε έχουν σχέση με θέματα εσωτερική ασφαλείας. Πήγαμε λοιπόν στον ΠΟΕ, όπω έκαναν και πολλοί συνάδελφοι και φίλοι, η Νορβηγία, ο Καναδάς, το Μεξικό, η Ιαπωνία και άλλε χώρες, τι οποίε ξεχνώ αυτή τη στιγμή. Επίσης θεσπίσαμε αντίμετρα, τα γνωρίζετε, δημοσιεύτηκαν και ετοιμαζόμαστε να δημοσιεύσουμε ο, κανονάς, ο κατάλογος με είναι στο Συμβούλιο αντίμετρα για τις θέσεις των ΗΠΑ όσον αφορά την αυτοκινητοβιομηχανία. Όλα αυτά που γίνονται επηρεάζουν όχι μόνο την παγκόσμια οικονομία αλλά και τι ΙΠΑ Έχουν επιπτώσει στο εσωτερικό των ΙΠΑ και πολλέ εταιρείε τη και πολλοί πολιτικοί μάλιστα και πολλοί άλλοι εκφράζουν ανοιχτά τις ανησυχίες τους γιατί πολλά πράγματα είναι πιο ακριβά πλέον στη ΣΥΠΑ. Οι δεσμοί το ξέρουμε όλοι. Είναι κάτι κακό. Επίσης δεν συμφωνούμε με όλου τους δεσμούς που επέβαλαν η ΙΠΑ στην Κίνα. Και δεν είναι μόνο δεσμοί, είναι και άλλα πράγματα. Ε, γίνονται πράγματα από τη ΣΥΠΑ που δεν είναι σύμβατα με τον ΠΟΕ. Πρόκειται για εμπορικό πόλεμο. Οι Αμερικανοί επιδοτούν κάποιες βιομηχανίες τους. Υπάρχει περιβατισμός από το κράτος, έχουμε θέματα μεταφορά τεχνολογίας, όλα αυτά να καταθέσουμε στον ΠΟΕ, όχι μόνο εμείς, αλλά και άλλοι, στην προσπάθεια μετατροπής του ΠΟΕ σε έναν καλύτερο ΠΟΕ και για να βελτιωθεί και η Κίνα. Λοιπόν, συνεργαζόμαστε με τις ΗΠΑ, αλλά δεν συμφωνούμε προφανώς με τη θέση τους. Ε, με την επιβολή τεράστιων δασμών εις βάρος της Κίνας ή της Τουρκίας. Λοιπόν, έχουμε διαφωνίε, διαφωνίες, επαναλαμβάνουμε τι είπα, σε όλα τα μέτωπα. Όμω, πιστεύουμε ταυτόχρονα ότι αν υπάρχει έστω κάποια δυνατότητα να βρούμε κάποια κοινά σημεία, έστω λίγα, να ξεκινήσουμε από κάπου για να βρούμε λύσει. αυτό θα είναι καλό. Στο ταξίδι του πρόεδρου Γιούνκερ πήγε, ξέρετε, στο Λευκό Οίκο. Αυτά έγιναν το καλοκαίρι. Τα συζητήσαμε όμω και με τα κρατη και μετά έχουμε την εντολή τη Σόφια. Αν θυμάστε, θυμηθείτε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τη Σόφια. Υπάρχει εντολή λοιπόν για την Κομισιόν. Τι κάναμε λοιπόν μετά, δημιουργήσαμε μια ομάδα εργασία. Δεν χρειαζόμαστε εντολή γι' αυτό, για να δημιουργήσουμε μια ομάδα εργασία και είπαμε ότι θα ξεκινήσουμε από το να διερευνήσουμε πώ περίπου θα χειριστούμε το θέμα. Δεν ξεκινούμε ξανά συνομιλίε για την TTIP δεν αναβιώνουμε την TTIP και υπάρχουν πολλοί λόγοι γι' αυτό. Αναφέρεται ορισμένους από αυτούς. Η TTIP λοιπόν δεν είναι στο τραπέζι. Πρόκειται για κάτι πιο περιορισμένο, ενδεχομένω να είναι μια πιο μικρή εμπορική συμφωνία που φέρα μόνο τους δασμούς σε προϊόντα, σε εμπορεύματα. Θέλαμε κάτι περισσότερο και εμείς και είπα, αλλά και αρχίζουν οι δυσκολίες. Γι' αυτό λέω ας ασχοληθούμε με τους δεσμούς και μόνο πρώτα απ' όλα. Ιδανικά θα θέλαμε να περιορίσουμε τους δεσμούς, όλους τους δεσμούς στο μηδέν. Αμοιβαίως. Και αν το πετύχουμε αυτό θα είναι καλό και για εμάς και για τις είπα. Παντού δασμοί μηδέν. Θα το κάνουμε αν το κάνουν και αυτοί. Αλλά θα δούμε τι θα πράξουν οι Αμερικανοί. Στο πλαίσιο αυτό, και αυτό ο είπα στις συμφωνίες τους θέλουν και την άδεια εξαγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου. Το αν θα αγοράσετε ή όχι, δεν θα σα το πει η Κομισιόν, αλλά ξέρω ότι κάποια κρατημέλη θα ήθελαν να αγοράζουν υγροποιημένο φυσικό αέριο από τι ΗΠΑ. Αν το θέλουν, να το κάνουν. Και εμεί θα προσπαθήσουμε να διευκολύνουμε αυτή τη διαδικασία. Οι υποδομέ υπάρχουν σε κάποιε χώρε. Το θέμα είναι, να δούμε λοιπόν από εδώ και πέρα, μπορούμε να περιδιαγράψουμε υπογράψουμε μια περιορισμένη, πεπερασμένη εμπορική συμφωνία για τους δασμούς. Αν ξεκινήσουμε από εκεί και πετύχουμε, ε, του ενδιαφέρει η γεωργία, μα ενδιαφέρουν οι δημοσίες συμβάσει κλπ. Εμεί δεν θέλουμε την γεωργία για πολλούς λόγους, του είπατε κι εσεί. Εάν, επαναλαμβάνω, μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι αυτό είναι το πεδίο, το αντικείμενο μιας συμφωνίας, τότε θα πάμε στο Συμβούλιο και θα ζητήσουμε μια εντολή. Γιατί το ξαναλέω. Δεν έχουμε ξεκινήσει καμία διαπραγμάτευση. Δεν υπάρχει αντικείμενο. Πρώτα πρέπει να ερεμήσουμε, να υπάρξει αποκλιμάκωση τη κατάσταση και μετά θα δούμε. Ο πρόεδρο Γιούνκερ και εγώ στείλαμε το μήνυμα ότι θέλουμε η ΕΠΑ να καθίσει στο τραπέζι με τρόπο θετικό και να ξεκινήσουμε από την κατάργηση των δασμών για το χάλιβα και το αλουμίνιο. Θα δούμε που θα πάει όμω αυτό. Συνεχίζουμε να πιστεύουμε ότι η δεσμή αυτή είναι παραδεκτοί. Οι ΙΠΑ υποσχέθηκαν ότι στο πλαίσιο αυτών των συνομιλιών δεν θα επιβάλλουν εν μεταξύ ε, ούτε δασμού ούτε ποσοστό. Αν γίνει κάτι τέτοιο, εμεί θα αποχωρήσουμε αμέσω από τι διαπραγματεύσει. Και ότι οι δεσμοί, η ποσοστό για τα αυτοκίνητα δεν είναι καλή για την εκλογική σα περιφέρεια. Τώρα για τα πρότυπα και του κανονισμού. Εδώ έχει γίνει πολύ σημαντική δουλειά στο πλαίσιο της TTIP, να ξέρετε, και υποστηρίζουμε την ίδια θέση. Είχαμε θέματα εξοπλισμού, αυτοκινήτων, θέματα ασφάλειας κλπ. Αυτά χρειάστηκε να γίνουν και μία και δύο φορές. Αλλά κάποια στιγμή πρέπει να αναγνωρίσουμε αμοιβαίως τα πρότυπα και τα πλαίσια της TTIP έχει γίνει προεργασία. Αυτό θα είναι καλό για όλους. Και πάλι, σε καμία περίπτωση δεν θα αποδεχθούμε ταπείνωση των δικών μας προτύπων. Δεν πρόκειται να γίνει αυτό σε καμία περίπτωση. Πρέπει να με πιστέψετε. Αν έχετε παράδειγμα, να μου το πείτε παρακαλώ. Άρα, εκεί δεν υποχωρούμε. Ούτε ξεκίνησαμε να συζητάμε γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς που είναι πηγή ανησυχίας. Από εκεί πέρα κάποια θέματα θα τα χειριστείτε εθελοντικά, σε θελουσία βάση, πάντως μας αφορούν όλους. Επίσης, θα προσπαθήσουμε μαζί με τη ΣΥΠΑ να μεταρρυθμίσουμε τον ΠΟΕ. Σε κάποια θέματα συμφωνούμε. Για το εφετείο ξέρετε ότι διαφωνούμε και είμαστε σε τέλμα αυτήν την στιγμή. Δεν έχουμε ξεβριλήσει, αλλά δεν θα καταλήψουμε και τις προσπάθειες. Δεν έχουμε λοιπόν ξεκινήσει διαπραγματεύσεις. Δεν έχουμε κάνει παραχωρήσεις κύριε Σιγητά. Προσπαθούμε ακόμη να δούμε αν υπάρχει κοινό τόπος για κάποιες πρώτες προσπάθειες. Αυτό κάνουμε αυτή τη στιγμή. Για τη σόγια. Εισάγουμε όλο και περισσότερους σπόρους σόγιας από τη ΣΥΠΑ. Γιατί? Λόγω δοσμολογικού πολέμου μεταξύ ΙΠΑ και Κίνας. Η Κίνα αγοράζει σόγια, όχι από τη ΣΥΠΑ αλλά από την Βραζιλία, το οποίο σημαίνει ότι η Βραζιλία δεν μπορεί να μας πουλήσει όση σόγια θα θέλαμε. Και εμείς δεν παράγουμε αρκετή σόγια στην Ευρώπη, παράγουμε στην Ιταλία, αλλά δεν είναι αρκετή, είναι κυρίω για ζωοτροφέ. Οπότε που θα στραφούμε αναγκαστικά στη ΣΥΠΑ. Η ΙΠΑ παράγει πάρα πολύ σόγια και γι' αυτό εισάγουμε σόγια από τη ΣΥΠΑ. Είμαστε μια ελεύθερη οικονομία. Δεν λέμε σε κάποιον τι θα κάνει, από πού θα εισαγάγει ή από πού δεν θα εισαγάγει. Ο κόσμος στρέφεται προς τη ΣΥΠΑ αναγκαστικά. Και γι' αυτό τον λόγο οι σπόροι αυτοί που είναι εγκεκριμένοι εισάγονται σε πολύ μεγάλες ποσότητες από τις ΕΠΑ. Είναι εγκεκριμένοι από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφαλής Τροφίμων. Η, αγορά είναι ελεύθερη ε, και οι επιχειρήσεις εισάγουν ελεύθερα από τις υπενγκεκριμένους πόρους. Αυτά για τη σόγια. Τι ξεχνάω. Αυτά ως προς τις διαπραγματεύσεις. Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, δεν είναι σαφές σε καμία περίπτωση. Θα προσπαθήσουμε να οριστικοποιήσουμε το χρονοδιάγραμμα κατά τη διάρκεια της παρούσας θητείας της Κομισιόν και να προχωρήσουμε και τις διαπραγματεύσεις, αλλά αυτό εξαρτάται και από το Συμβούλιο. Θα το κρατήσουμε ενήμερο. Εννοείται σε κάθε περίπτωση. Το Buy American, τον νόμο Buy American, το βρίσκουμε παράδεκτο. Θέλουμε γι' αυτό να εντάξουμε και τις δημόσιες συμβάσεις στις ομιλίας. Νομίζω δεν είναι δυνατόν προς το παρόν, αλλά θα δούμε. Βιώσιμη ανάπτυξη κλπ. Αυτά κοιτάξτε, δεν... είναι εκτός και της ε, εννοείται ότι σε κάθε περίπτωση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμμετέχει στη διαδικασία, γι' αυτό είμαι και εδώ. Θα συνεχίσουμε σήμερα και οποτεδήποτε άλλοτε χρειαστεί. Θα χρειαστούμε εντολή, εννοείται, το επαναλαμβάνω, όταν ξεκινήσουμε τι διαπραγματεύσει και εννοείται ότι στις διαπραγματεύσει θα εμπλακεί και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τώρα, επειδή με ρωτήσετε, αλλάξαμε εμπορική πολιτική. Βεβαίω, αλλάξαμε εμπορική πολιτική. Είμαστε πιο διαφανεί, έχουμε ενσωματώσει τι αξίε μα, τονίζουμε τι αξίε μα, είμαστε πιο αποτελεσματικοί και εννοείται στη διαδικασία. Αυτή θα συμμετάσχει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Προβλέπετε και θα γίνει. Όταν λοιπόν ξεκινήσουμε, ε, οι συνομιλήσει θα είναι μεταξύ εμού ε, και του μονίμου αντιπροσώπου των είπα. Ο κ. Σελμάγερ προετοίμασε την συνάντηση μεταξύ των δύο προέδρων. Αυτή είναι, αυτός είναι ο ρόλος του. Συνεργάστηκε με συνεργάτες του πρόεδρου Τραμπ. Προετοίμασε πολύ ικανοποιητικά νομίζω αυτή την συνάντηση, η οποία έγινε σε επικοδομητική ατμόσφαιρα. Πήγε πολύ καλύτερα από ό,τι περιμέναμε. Από εκεί πέρα όμως σας είπα ποιοι ε, μεταξύ ποιων θα γίνουν οι διαπραγματεύσει. Κάποια στιγμή θα ανέβουμε και στο επίπεδο του Προέδρου και του Γραφείου του με τον Λευκό Οίκο. Πρόκειται για μια, θα πρόκειται για μια ευρύτερη εμπορική συμφωνία. Εφόσον δούμε ότι μπορούμε πραγματικά να προχωρήσουμε κάπως. Και για τον Καναδά, πιστεύω ότι πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι γίνεται με την ναύτα. Το Μέξικο και ο Καναδά συμφώνησαν. Η ε, κυρία Φίλαν, η Καναδή διαπραγματεύτρια είναι στις... Είπα στην Ουάσιγκτον, δεν θα υπογράψει ελευκό Είχαμε, είχαν πει κάτι για τον Αύγουστο, αλλά μα μένουν μόνο δύο ημέρε. Θα χρειαστεί λοιπόν περισσότερο χρόνο. δεν τελειώσουμε τον Αύγουστο και θα δούμε τι επιπτώσει θα έχει ναύτα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ΣΕΤΑ, ε, με τη ΣΕΤΑ κλείνουμε ήδη ένα χρόνο, πολύ σύντομα. Νομίζω ότι πήγαμε πολύ καλά. Οι Καναδοί την <laughs> αγαπούν. Δεν θα κάνουν τίποτα στην ναύτα που να δημιουργεί προβλήματα στην ΣΕΤΑ αλλά αυτό θα το επιβεβαιώσουμε όταν έχουμε μια σαφέστερη εικόνα της κατάστασης. Και για το δικό μας εμπορικό πλεόνασμα εις βάρος τον είπα. Κοιτάξτε, αυτό μπορεί να το μετρήσει κανείς με διαφορετικούς τρόπους. Δεν σύμφωνα αναγκαστικά με τον ορισμό του πρόεδρου Τραμπ. Μπορεί να το μετρήσει κανείς με διαφορετικούς τρόπους. στα προϊόντα έχουν πλεόνασμα, έχουμε μάλλον πλεόνασμα, στις υπηρεσίες είναι το αντίθετο. Αυτό εξαρτάται από τι αποταμιεύσει, τι καταναλωτικέ συνήθειε κλπ. Δεν υπολογίζονται όλα αυτά, ξέρετε, με τον ίδιο τρόπο. Οπότε δεν έχω και σχόλιο για την ε, γερμανική οικονομία. Η Κομισιόν διατυπώνει τα σχόλιά τη κάθε εξάμεινο στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Περιτεύει λοιπόν ε, και παρέλκει να σχολιάσω συγκεκριμένα κράτη-μέλη. Αυτά λοιπόν ελπίζω να τα ξεκαθάρισα, γιατί υπήρχαν πολλέ παρεξηγήσει και φόβοι. Ελπίζω να ε, διευκρίνησα την κατάσταση. Ευχαριστώ πολύ, Επίτροπε. Ναι, θέλω να ξαναπάρω το λόγο, παρακαλώ. Α, ναι, για τις βρώσιμες ελιές. Το συζητήσαμε και με τον κύριο Λαϊτάιζερ και με τον ε, κύριο Γκρός, ε, με πολλούς υπουργούς ε, το συζητήσαμε το θέμα αυτό και με τον Επιτροπό και ο Επιτροπός Χόγκαν επίσης το συζητάει. Είμαστε και σε στενή επαφή με την Ισπανική κυβέρνηση έτσι ώστε να δούμε πώς μπορούμε να υποστηρίξουμε την Ισπανική κυβέρνηση σε αυτό το θέμα. Θα συνεχίσουμε να το υποβάλουμε, να το αναφέρουμε στις παράλληλες συζητήσεις ως ε, εισηγητής αρμόδιος για τις σχέσεις ε, Ένωσης είπα να κάνω κάποιες τελικές παρατηρήσεις. Ευχαριστώ καταρχήν την Επίτροπο Μάλμστρομ που ήρθε και μας ενημέρωσε γρήγορα μετά τις συνομιλίες στην Ουάσιγκτον. Βλέπω ότι την προσέγγιση που ακολουθήσατε την ε, υποστηρίζετε Βεβαίω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα παρακολουθήσει τις εξελίξεις. Παρακολουθούμε με κριτικό πνεύμα. Η στρατηγική εμπόριο για όλους του 2015 είναι η κοινή βάση για την εμπορική πολιτική, θυμίζω. Και πάνω σε αυτή τη βάση γίνονται διαπραγματεύσεις και με άλλες χώρες ε, στον κόσμο. Και από ό,τι ακούσα και από άλλες χώρες είναι ότι εξεπλάγει λίγο εξεπλάγησαν λίγο για το γεγονός ότι ε, δεν καλύψαμε όλα τα θέματα στις συνομιλίες ε, με τις ΗΠΑ. Ε, τώρα διαπραγματευόμαστε με έναν ισχυρό εταίρο και δεν πρέπει να παραιτηθούμε όμως από τις αρχές μας. Αυτό να είναι σαφές. Και είμαι πεπισμένος και εν ώψη των παγκόσμιων αλλαγών που διαπιστώνουμε ότι ως Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ε, συμφωνούμε με την πολιτική του Διέρη και Βασίλευε. Αντίθετα πρέπει να προβάλλουμε ξεκάθαρα τις δικές μας θέσεις. Όλες αυτές οι εξελίξεις θα τις παρακολουθήσει από κοντά το Κοινοβούλιο και όταν φτάσουμε σε εντολή θα συζητήσουμε για αυτή τη διαπραγματευτική εντολή. Και το Κοινοβούλιο θα αποφανθεί σχετικά με τη συμφωνία. Θα θυμάστε ότι έχει ε, τύχει να απορρίψουμε εμπορική συμφωνία αν δεν την εγκρίνουμε. Ευχαριστώ για το διάλογο και ε, κλείνω το σημείο αυτό της ημερησίας διάταξης. Δύο θέματα ακόμα. Τα διάφορα, το 24, το αγαπημένο μου. Υπάρχει τίποτε. Ο κύριος Στάρτμορ. Είναι 11 και 53 και αν δεν κάνω λάθος, μέχρι τις 12.30 έχουμε διερμηνία. Έτσι δεν είναι. Έτσι δεν έλεγε και η ενημέρωση. μέχρι τις 12, 12 και 30, εντάξει. Πολλοί συναδελφοί ε, θα είχαν πράγματα να ρωτήσουν την Επίτροπο, αλλά υπήρχαν χρονικοί περιορισμοί. Καλό θα ήταν να ακούσουμε τους συναδέλφους για περισσότερο χρόνο. Καλό θα ήταν να έχουμε τη δυνατότητα και μεταξύ μας να συζητήσουμε, γιατί βεβαίως έχει άλλα καθήκοντα η Επίτροπος. Αλλά να σχολιάσουμε τα όσα είπε. Έχουμε 36 λεπτά. Μην τα σπαταλήσουμε και τα χάσουμε. Χθες είχαμε μία μελέτη 55 σελίδων ε, από την ΑΦΕΤ και από την δική σας ε, επιτροπή από κοινού έκθεση και οι συνάδελφοι και εγώ περιοριστήκαμε στα δύο λεπτά μόνο. Καταλαβαίνω ότι όλοι είναι απασχολημένοι τις χρονικές πιέσεις Βεβαίως και οι διερμηνείς κάνουν καλή δουλειά και... Ε, αλλά δεν αξιοποιούμε με το βέλτιστο τρόπο την υποδομή που έχουμε. Ιδιαίτερα σήμερα ισχύει αυτό. Α, δεν συμφωνώ. Εμείς το χρόνο μας τον αξιοποιούμε καλά και ε, αρχίσαμε μάλιστα και μισή ώρα νωρίτερα χθε το απόγευμα για να τα προλάβουμε όλα. Διαδικαστικά. Πρόταση κάνω. Ευχαριστώ την Επίτροπο που έχει φύγει βέβαια και να προτείνω να κάνουμε μια συζήτηση μεταξύ μας κάποια στιγμή σχετικά με, τα, με αυτά που είπε η Επίτροπος. Πρόεδρος, ε, έχουμε μια επιτροπή παρακολούθησης για τη ΣΥΠΑ. Θα κάνουμε συζήτηση σε βάθος στα, ε, εκεί. Και αυτό θα γίνει σύντομα. Τελειώσαμε και το 24-25 προσεχή συνεδρίαση 27 Σεπτεμβρίου στις Βρυξέλλες. Ε, ευχαριστώ πολύ.